Καλησπέρα σε αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πρέπει να ξεκινήσουμε αμέσως. Παρακαλώ καθίστε. Allora, Θα δώσω το λόγο στον καθηγητή Βάιλερ, που είναι αυτή τη στιγμή διευθυντής του κέντρου Ζαμονέ για, τα, για την περιφερειακή οικονομία στο School Law. Ε, τέλεσε καθηγητής σε πολλά πανεπιστήμια και στο Collège Rop και είναι καθηγητής ε, ε, διεθνούς δικαίου και γράφει και, στο, και στη βιβλιογραφία για θέματα διεθνούς δικαίου. Παρακαλώ τον καθηγητή Βάιλερ να λάβει θέση.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 Σας δίνω το λόγο καθηγητά Βάιλερ και σας ευχαριστούμε ε, θερμά για την παρουσία σας. Θα ακούσουμε λοιπόν την παρέμβαση του καθηγητού Βάιλερ. Το θέλουμε παρακαλώ να μην ξεπεράσει τα 15 λεπτά. Ευχαριστώ. Το θέμα μας εδώ πέρα είναι η σχέση μεταξύ ατόμου και της Ένωσης και συχνά αυτό εκφράζεται υπό την έννοια της ε, νομοποίησης η οποία νομοποίηση συχνά συγχέεται με την δημοτικότητα αλλά σε περίοδους κρίσης ισχύει το αντίστροφο και καιρούς κρίσης ε, χρειάζονται αντιδημοφιλή μέτρα ε, με τα οποία συχνά δεν συμφωνεί ε, ο λαός ή δεν στηρίζει άμεσα. Και ακριβώς σε αυτές τις συνθήκες κρίσης η νομιμότητα της πολιτείας, της διακυβέρνησης ακριβώς δοκιμάζεται γιατί αν υπάρχει βαθιά νομοποίηση μπορούν να ληφθούν μη δημοφιλή μέτρα τα οποία θεωρούνται όμως νομοποιημένα. Η θέση μου λοιπόν εδώ πέρα θα είναι πως στην κρίση αυτή έχουν εξαντληθεί οι πόροι νομοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο μηδέν και αυτό εμποδίζει την Ένωση από το να αναλάβει αποφασιστική δράση και την αναγκάζει να βασίζεται στα αποθέματα νομοποίησης των κρατών μελών. Το να αντιληφθούμε λοιπόν αυτή την εξάντληση των αποθεμάτων νομοποίησης της Ένωσης είναι σημαντικό εάν μέσω μακροπρόθεσμα ε, σχηματιστεί ε, ένας διαφορετικός σχηματισμός για να αποφευθούν αυτά στο μέλλον. Οπότε, το πρώτο το οποίο πρέπει να ρωτηθούμε είναι γιατί λέω πως έχουν εξαντληθεί οι πόροι αυτοί της νομότας και δεν έχει την νομότητα αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει και μια κυβέρνηση σε καιρούς κρίσης για να μπορεί να δράσει με τρόπο μη δημοφιλή αλλά να θεωρείται ε, Έχουμε λοιπόν στην πολιτική επιστήμη τριών ειδών νομοποίηση. Έχουμε την νομοποίηση της ε, διαδικασίας τη δημοκρατία δηλαδή θα λέγαμε και την νομοποίηση των αποτελεσμάτων και μετά βεβαίως υπάρχει και η διαδικασία του σκοπού καμιά φορά αυτό λέγεται και πολιτικός μεσιανισμός το όνειρο το οποίο, το όραμα το οποίο έχει κανείς θα ήθελα λοιπόν να εξηγήσω σύντομα γιατί ο πολιτικός μηχανισμός και η νομοποίηση του αποτελέσματος δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωσή μα και μετά να αφιερωθώ λίγο στην ε, νομοποίηση της διαδικασίας. Εδώ και δεκαετίες, είτε ανοιχτά είτε σιωπηλά, η πηγή της νομοποίησης ήταν τα αποτελέσματα. Όταν υπήρχαν αποτελέσματα ήταν ε, νομοποιημένοι και ο καλύτερος τρόπος να νομοποιηθεί ένας πόλεμος βεβαίως είναι να τον ε, κερδίσει κανείς. Αυτές είναι οι λειτουργικές οι λεγόμενες θεωρίες όταν και στη διακήρυξη Σουμάν μιλούσαν για μια de facto αλληλεγγύη και συγκεκριμένα επιτεύγματα. Δηλαδή όταν υπάρχουν αποτελέσματα και προφανώς σε καιρούς κρίσης όπως σήμερα δεν μπορούμε να βασιστούμε σε αυτό. Δεν έχει σημασία εάν η κρίση οφείλεται στην Ένωση ή όχι ή αν οφείλεται στην Κομισιόν ή στο Συμβούλιο ή όχι. Σημασία έχει το πώς το βλέπει ο λαός και ο λαός θεωρεί πως στην περίοδο αυτή η Ένωση δεν παράγει αποτελέσματα. Αντιθέτω, μάλιστα δημιουργεί το πρόβλημα. Όπω είπα, δεν έχει σημασία αν ισχύει αυτό στην πραγματικότητα. Αυτή είναι η ιδέα, η αντίληψη. Αν δούμε διάφορες ε, δημοσκοπήσεις. Οπότε δεν έχουμε αυτή τη στιγμή την νομοποίηση, όπως είπα, του από το αποτέλεσμα. Ο πολιτικός μεσιανισμός λοιπόν, το όνειρο της Ευρώπης ήταν ο ισχυρότερος νομοποιητικός παράγοντας στην ε, ιστορία της Ένωσης. Εάν πάμε στην περιφερειακή βάση, ε, μην ξεχνά πως αρχικά το Κοινοβούλιο ήταν μια συνέλευση, δεν είχε καθόλου ε, αρμοδιότητες, ήταν κάποιοι αξιωματούχοι των κρατών μελών και κάποια άλλες επιτροπές και δεν υπήρχαν αποτελέσματα. Ήταν ακόμα στην πολύ αρχή και όμως ήταν πάρα πολύ νομοποιημένο γιατί υπήρχε ένα όνειρο. Υπήρχε το όνειρο του Σούμαν, το όνειρο του να γίνουν τα, ε, τα ξύφη άρωτρα όπως έλεγαν από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και να υπάρξει ένα ε, καλύτερο μέλλον. Και ήταν κάτι το οποίο συνάρπαζε. Γι' αυτό το βάζω στην κατηγορία του πολιτικού μεσιανισμού. Δεν έχει σημασία αν τα μέσα δεν ανταποκρίνονταν στις συνήθειές μας, στις συνήθειες περί δημοκρατικής διακυβέρνησης, καθώς ήταν ένα συναρπαστικό όνειρο στο όνομα το οποίο μπορούσαν να επιτευχθούν πάρα πολλά και ο κόσμος ήταν διατεθειμένος να κάνει και θυσίες και να δεχτεί αυτό το οποίο έκανε η Ένωση γιατί πήγαινε προς αυτό το συναρπαστικό όνειρο. Αυτό δεν μπορεί να κρατήσει. Ο πολιτικός μεσιανισμός πάντα καταραίει. Για δύο λόγους. Πρώτον, εάν ε, ε, επιτύχει, γιατί αυτή τη στιγμή ε, πραγματοποιηθεί το όνειρο, δεν είναι πλέον όνειρο, οπότε δεν υπάρχει κάποια προσδοκία. Και πιο συχνά η η υλοποίηση του ονείρου βεβαίως δεν ανταποκρίνεται σε αυτό, ποτέ σε αυτό το οποίο ήταν το όνειρο γιατί αντιλαμβάνεστε ο γάμος όπως λένε ποτέ δεν είναι σαν το μήνα του μέλητος όταν φτάνει κανείς στη γη της επαγγελίας είναι τελείως διαφορετική από αυτό το οποίο φανταζόταν το ίδιο και με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση αν θέλετε να κάνουμε μια παρομοίωση αν συγκρίνουμε τις 800 λέξεις της διακήρυξης Σουμάν με τις 130.000 λέξεις της συνθήκης της Λισαβόνας αντιλαμβάνεστε την διαφορά ανάμεσα στο όνειρο και την πραγματικότητα. Οπότε είναι δύσκολο να διατηρηθεί αυτός ο πολιτικός μεσιανισμός. Αλλά θα πω και κάτι άλλο. Τώρα που η Ευρώπη ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη, έχει επιτύχει τον στόχο της μακροπρόθεσμης ειρήνης, θυμάμαι όταν ο Μιτεράν και ο Κόλ είχαν εμφανιστεί στην τηλεόραση και προσπάθησαν να πείσουν ε, τους Γάλλους να υπερψηφίσουν τη συνθήκη του Μάστριχτ μιλούσαν για την ιστορική συμφιλίωση μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας και οποιοδήποτε ήταν κάτω των 45 δεν καταλάβαινε τι εννοούσαν. Αυτό είναι σημάδι της επιτυχίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Το πρόβλημα λοιπόν είναι τώρα να βρούμε ένα νέο όραμα, μια νέα μορφή πολιτικού μεσιανισμού κάτι το οποίο δηλαδή μπορεί να σαγηνεύσει πραγματικά. Δεν το έχουμε τώρα αυτό. Το να λέμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερη πολιτική ένωση για να σωθεί το ευρώ είναι περισσότερο ένα πικρό φάρμακο το οποίο μας ε, καταπιέζουν να καταπιούμε γιατί αλλιώς θα αποτύχει η Ευρώπη. Δεν είναι κάτι το συναρπαστικό. Οπότε δεν υπάρχει κάτι που να υποκαταστήσει τον αρχικό πολιτικό μεσιανισμό που ήταν ο κινητήρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε, έρχομαι τώρα στη δημοκρατία. Και εδώ πέρα υπάρχει ένα παράδοξο. Ποιο είναι αυτό. Το δε, το δε αυτή την παρουσίασή μου τη λέω «Δημοκρατία χωρίς το λαό». Βλέπουμε εδώ πέρα πως ε, οι αρχές της δημοκρατίας γίνονται σεβαστές. Υπάρχει ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχει περισσότερες ε, εξουσίες, είναι συνομοθέτης, εκλέγεται δημοκρατικά. Οπότε το ερώτημα είναι <clears throat> πού είναι το δημοκρατικό έλλειμμα και όμως ας δούμε λίγο το παράδοξο. Θυμάμαι το 1979 στι πρώτε άμεσε εκλογέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπήρχε μια απογοήτευση για το ότι η προσέλευση ήταν χαμηλή. Και δεν το συγκρίνουμε βεβαίω με τι ΗΠΑ που είναι πάντα χαμηλή η προσέλευση, το συγκρίναμε με τι εθνικέ εκλογέ των κρατών μελών. Και ήταν πολύ χαμηλή η προσέλευση. Και πάρα πολλοί τότε και εγώ είπαν πω δεν ε, πρέπει να προκαλεί εντύπωση γιατί έχει ελάχιστε εξουσίε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί να πάει κανεί να ψηφίσει. Και η πρόβλεψη ήταν πω όταν θα είχε αρμοδιότητε θα ε, πήγαινε ο κόσμο να ψηφίσει. Όταν θα φαινόταν πω έχει κάποια ουσιαστική εξουσία η προσέλευση θα αυξανόταν. Και συνέβη το αντίθετο. Με κάθε διακυβερνητική διάσκεψη απέκτησε περισσότερες εξουσίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οπότε σήμερα είναι πραγματικά συνομοθέτης μαζί με το Συμβούλιο των Υπουργών. Και αν δούμε όμως την προσέλευση στις ευρωεκλογές, υπάρχει σταθερή μείωση. Αυτό είναι το παράδοξο. Περισσότερες εξουσίες, λιγότερη εμπλοκή των πολιτών, λιγότερη εμπιστοσύνη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τουλάχιστον όπως τη μετράμε από το ποσοστό των ανθρώπων που κατεβαίνουν να ψηφίσουν. Αυτό είναι βασικό για να αντιληφθούμε τα δημοκρατικά προβλήματα της Ευρώπης. Πώς θα εξηγούμε λοιπόν αυτά. Θα ήθελα λοιπόν ε, εγώ να ε, πρόσφερω κάποιες εξηγήσεις. Πρώτον, έχουμε στα κράτη-μέλη διαφορετικά δημοκρατικά συστήματα. Το, δημοκρατικό, το προεδρικό σύστημα της Γαλλίας διαφέρει πολύ από το κοινοβουλευτικό σύστημα της Αγγλίας και το Βρετανικό διαφέρει από το Γερμανικό και το Ιταλικό. Εγώ όμως θα ήθελα να αναφέρω δύο αρχές που ισχύουν σε όλες τις δημοκρατίες στην Ευρώπη. Δεν καθορίζουν το τι είναι δημοκρατία, αλλά εάν δεν υπάρχουν, δύσκολα μιλάμε για δημοκρατία. Δεν σημαίνει πως αν τα έχει κανείς έχει και δημοκρατία αυτομάτως, αλλά εάν δεν τα έχει, δεν έχει. Το πρώτο είναι η αρχή της εκπροσώπησης. Εάν αρκετοί άνθρωποι πάνε να ψηφίσουν με κάποιον τρόπο, αυτό πρέπει να αντικατοπτρίζει τις ε, προτιμήσεις ε, του νομοθετικού σώματος ε, και της διοίκησης. Έχει διαφορά αν βγει Ρόμνη ή Ομπάμα, αν είναι Μέιτζορ ή Τόνι Μπλερ, αν είναι ο Ολάντ ή ο Σαρκοζή. Ίσως όχι τεράστια διαφορά, αλλά έχει διαφορά σε πολιτικές αναδιανεμητικές, εξωτερική πολιτική κτλ. Οπότε οι προτιμήσεις του ψηφοφόρου μεταφράζονται σε πολιτική και διακυβέρνηση. Και αυτό στην Ευρώπη δεν ισχύει. Δηλαδή η σχέση μεταξύ προτίμησης του ψηφοφόρου και αποτελέσματος είναι πάρα πολύ ασθενής. Δεν έχει σημασία αν είναι κέντρο αριστερή ή κέντρο δεξιά η πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν βλέπουμε να μεταφράζεται αυτό στην πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κάτι διαφορετικό. Η πιο θεμελιώδης αρχή της δημοκρατίας είναι η αρχή της εκπροσώπησης, όπου ο ψηφοφόρος ξέρει πως εάν ψηφίσουν αρκετοί σαν και εμένα θα επηρεάσουμε το τι κάνει η Ένωση. Αυτό δεν συμβαίνει. Αυτό φαίνεται στα ε, εκλογικά προγράμματα των κομμάτων. Δεν παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που είναι διαφορετικό από τους άλλους. Όλοι είναι υπέρ ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κλασικά εκεί πέρα, αλλά δεν έχει κανείς την αίσθηση πως ψηφίζει ένα πρόγραμμα και έχει διαφορά εάν ψηφίσει τους σοσιαλιστές ή τους σοσιαλδημοκράτες, πως θα αλλάξει η Ευρώπη. Ε αυτό σχετίζεται με τη σχέση μεταξύ Κοινοβουλίου και Κομισιόν. Η Κομισιόν είναι περήφανη για το ότι δεν είναι κομματικοποιημένη. Δεν είναι σωστό να είναι κανείς ε, υπέρ ενός κόμματος στην Κομισιόν. Οπότε κάποιος το είχε πει ε, πριν από πολλά χρόνια και ισχύει. Δεν είναι τόσο δημοκρατικό έλλειμμα, αλλά πολιτικό έλλειμμα. Και δημοκρατία χωρίς πολιτική δεν είναι δημοκρατία. Και δεν υπάρχει ακριβώς αυτή η ζωτική λειτουργία της δημοκρατίας, ότι οι προτιμήσεις δηλαδή μεταφράζονται σε πολιτική. Δηλαδή και να έχει εξουσία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί να πάω να ψηφίσω άμα δεν κάνει διαφορά. Πρέπει, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Αυτή είναι η αλήθεια. Και το δεύτερο, κύριε Πρόεδρε, είναι η αρχή της λογοδοσίας. Οι Άγγλοι έχουν μία έκφραση που είναι διώχτε τα, καθάρματα. Δηλαδή έχουμε τη χύψη κυβέρνηση, δεν μας αρέσει ο Σαρκοζή και τον διώχνουμε και βγαίνει ο Ολάντ. Και μετά από 6, 7, 8 χρόνια μπορούμε και τα προηγούμενα καθάρματα να τα διώξουμε. Το διώχτετε τα καθάρματα δεν αφορά μόνο το νομοθετικό πρόγραμμα, αφορά και την απόδοση και το ότι δεν μ' αρέσει το, το πώς κυβέρνησαν αυτοί οι άνθρωποι είναι ζωτικό στοιχείο της δημοκρατίας. Σε καμία χώρα μας, σε όλες τις χώρες μας, υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξουμε την κυβέρνηση. Στην Ευρώπη έχουμε διακυβέρνηση, αλλά όχι κυβέρνηση. Οπότε η θεωρητική δυνατότητα της Κομισιόν να απολύσει την Κομισιόν δεν ισχύει, δεν ταυτίζεται με αυτό το οποίο λέμε αλλαγή κυβέρνησης. Γιατί η διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής, Κομισιό, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με είναι μεταξύ Κομισιών, Συμβουλίου, Κοινοβουλίου κτλ. Και αυτό είναι απλά ένα γεγονός. Δεν υπάρχει κάποια στιγμή στο χρονοδιάγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία εάν καταψηφίσουν οι πολίτες μπορούν να διώξουν τα καθάρματα. Δεν λειτουργεί έτσι το σύστημα και πάλι αρνούμαστε στους πολίτες ένα θεμελιώδες δικαίωμα και μια θεμελιώδη πτυχή της δημοκρατίας. Δεν γίνεται δηλαδή. Δεν του ψηφίζεις και πάλι οι ίδιες φάτσες είναι. Και ξέρω πως ο ψήφος μου δεν αλλάζει τίποτα. Ε, γιατί να πάω να ψηφίσω. Τι Vox Populi είναι αυτό. Αυτή μάλλον. Η φωνή του λαού. Δεν μιλάω τώρα για περιπτώσεις ε, υπεξαίρεσης ε, από πλευρά αξιωματούχων οι οποίοι πράγματι λογοδότησαν. Εγώ μιλάω για πολιτική λογοδοσία. Μπορεί κάποιος να μου πει ένα παράδειγμα από το 1979 και μετά, αλλά και πιο πίσω στο παρελθόν, όπου είχαμε πολιτική αποτυχία και κάποιος πλήρωσε πολιτικό τίμημα. Δεν επανεξελέγει και τα λοιπά δεν συμβαίνει για τους ευρωβουλευτές, δεν συμβαίνει για τα μέλη της Κομισιόν. Και ε, βλέπετε τι σημαίνει. Και υπήρχαν μεγάλες αποτυχίες. Η, η ατζέντα της Λισαβόνας, η λεγόμενη. Ε, δεν ήταν και επιτυχία. Η, η Κοπενχάγη και το φιάσκο εκεί πέρα. Ποιος πλήρωσε το πολιτικό τίμημα. Οπότε, όχι μόνο δεν μπορούμε να τα διώξουμε τα καθάρματα από πλευράς δομικής του συστήματος, αλλά δεν υπάρχει και πολιτική λογοδοσία. Οπότε, δεν πρέπει να μας προξενεί έκπληξη. Εάν αυτές οι δύο ε, βασικές εκφάνσεις της δημοκρατίας, δηλαδή η πολιτική εκπροσώπηση, η απόψη μου να μεταφράζω στην πολιτική και πολιτική λογοδοσία ότι αν ψηφίσουμε αρκετοί μπορούμε να τους διώξουμε, αν δεν υπάρχουν αυτά, δεν πρέπει να μας προξενεί η εντύπωση το ότι οι πολίτες Ευρώπης γυρνάνε την πλάτη τους και λένε οι ευρωεκλογέ δεν είναι αυτό το οποίο μας είχαν υποσχεθεί και ψάχνουν άλλους τρόπους βεβαίω για να εκφραστούν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό εξηγεί το παράδοξο το αρχικό. Αν έχω χρόνο, κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω κάτι ακόμα, αλλά μπορώ να σταματήσω εδώ πέρα, αν θέλετε. Ένα πράγμα θα πω ακόμα. Ξέρετε, όταν μιλάμε για δημοκρατία, η εργασία μου, όπως είπα, λέγεται δημοκρατία χωρίς το λαό. Γιατί εδώ πέρα έχουμε μια δομική αποξένωση του λαού, παρά το ότι το κοινοβούλιο έχει εξουσίες και ο κόσμος έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει, αλλά μας γυρνάνε την πλάτη. Ξέρετε, σε κάποια κράτη-μέλη είναι κατά από 30% η προσέλευση. Και αν δεν υπήρχαν και κάποιε χώρε που είναι υποχρεωτική η ψηφοφορία, θα έπεφτε συνολικά το ποσοστό κατά το 50%. Οπότε έχουμε αυτή τη μία έννοια με την οποία έχουμε δημοκρατία χωρίς το λαό, αλλά υπάρχει και άλλη μία έννοια. Όταν μιλάμε για δημοκρατία, ξέρετε τις ε, αρχαίες ελληνικές λέξεις, και βέβαια όταν μιλάμε για Δήμο μιλάμε για το λαό και όπω είχαν πει και οι Αμερικανοί είναι από τον λαό, για τον λαό, με τον λαό. Ένα από τα προβλήματα λοιπόν με την ευρωπαϊκή αυτή ε, υπηκότητα είναι ότι δεν υπάρχει η έννοια του Δήμου, δεν υπάρχει Ευρωπαϊκός Δήμος. Τα τελευταία 50 χρόνια ε, γράφει ο κόσμος πως δεν υπάρχει Ευρωπαϊκός Δήμος ε, και δεν μπορεί άρα να υπάρχει δημοκρατία. Όλα αυτά ένιωσαν ακαδημαϊκά μπλα μπλα. Τους άρεσαν δηλαδή οι κάποιους πανεπιστημιακούς η αρχαιοελληνική λέξη, εγώ το είχα γράψει αυτό πριν από 15 χρόνια και μου λέγανε «Μα τι είναι αυτά που λες τώρα». Τώρα όμως, στην κρίση του ευρώ, βλέπουμε ξεκάθαρα το πρόβλημα του ότι δεν υπάρχει δήμος και άρα δεν υπάρχει δημοκρατία. Και εξηγούμε. Γιατί όλοι ξέρουμε τι λύση στο ευρώ, χρειαζόμαστε κάποιο είδους δημοσιονομική ένωση. Δηλαδή όταν ε, φτιάχτηκε το ευρώ, θυμάμαι το Μάρτι Φέλσιν στο Χάρβαρτ, ε, ο οποίο χαιρετήσει τι θα γίνει με το πρώτο ασύμετρο σοκ όταν δεν υπάρχει ένα μηχανισμό για να μεταφέρει κονδύλια από την Καλιφόρνια α πούμε στη Βιρτζίνια ή το αντίστοιχο από τη Γερμανία στην Ελλάδα. Και ο Φέλτσιν το, το είχε πει ήδη από την αρχή. Τι θα γίνει σε αυτήν την περίπτωση. Χρειάζεται λοιπόν κάποια μορφή δημοσιονομική ένωση. Μπορεί να γίνει με διάφορου τρόπου, αλλά κυρίε και κύριοι, και κύριε Πρόεδρε, υπάρχει μια κοινωνική διάσταση στη Δημοσιονομική Ένωση. Η κοινωνική διάσταση σχετίζεται με αυτό το οποίο λέμε Δήμο και Δημοκρατία. Σα δώσω ένα παράδειγμα, γιατί χρησιμοποίησα τι ΗΠΑ. Α υποθέσουμε πως το Τέξα έχει δημοσιονομική κρίση όπως είχε με κάποιες ε, τράπεζες ε, στη δεκαετία του 90. Μια γελία ε, φούσκα κινήτων και χρεοκοπούσε η πολιτεία. Και υπήρχε μεγάλη συζήτηση Να τους γλιτώσουμε ή όχι να εξελασπώσουμε Νέα Υόρκη ή όχι. Η συζήτηση που έχουμε τώρα, να διασώσουμε την Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία. Το ενδιαφέρον σε αυτή τη συζήτηση ήταν πως κάποιοι λέγανε μην τους γλιτώστε. Ήτανε μοναταριστέ και τα λοιπά, να μάθουν έτσι την υπευθυνότητα, ηθικό κίνδυνο και τα λοιπά, τα έχετε ακούσει. Άλλοι έλεγαν όχι, όχι, όχι, εάν ε, δεν τους διασώσουμε το οικονομικό και κοινωνικό κόστος θα είναι υψηλότερο. Αλλά αυτό το οποίο δεν άκουσε κανείς ήταν γιατί εμείς στην Καλιφόρνια να ε, γλιτώσουμε τους Τεξανούς. Γιατί ήταν όλοι Αμερικάνοι. Και τα λεφτά. Ε, ήταν ομοσπονδιακά τα λεφτά της διάσωσης. Ήταν χρήματα τον είπα. Δεν έλεγε κανείς γιατί το Τέξας να διασώσει Καλά, αυτό μπορεί να το έλεγαν οι Τεξανοί, τέλος <laughs> πάντων. γιατί εμείς στη Μασαχουσέτη, ξέρω εγώ, να διασώσουμε τη Λουιζιάννα. Αυτό δηλαδή το ότι χωρίς Δήμο δεν υπάρχει δημοκρατία, το βλέπουμε τώρα. Γιατί ο λαός στη Γερμανία, στη Φιλανδία, στην Ολλανδία, που λένε μη διασώσουμε τους Έλληνες, δεν είναι γιατί είναι κατά της οικονομικής πτυχής. Δεν θέλουν να βοηθήσουν τους Έλληνες. Γιατί εμείς οι Γερμανοί να βοηθήσουμε τους Έλληνες, τους τεμπέληδες Ιταλούς ή τους Πορτογάλους και Δεν είναι ιδεολογική η αντίρρηση κατά της διάσωσης του μηχανισμού δεν βλέπουν την ανθρώπινη κοινωνική αλληλεγγύη με αυτό το λαό για να τον βοηθήσουν. Και ξαφνικά βλέπουμε πως το πρόβλημα εδώ πέρα δηλαδή η μη, ο μη ενιαίος δήμος που ήταν κάτι το ακαδημαϊκό, μια ακαδημαϊκή συζήτηση τώρα υπάρχει γιατί οι δυσκολίες που έχουμε για να βρεθεί μια λύση είναι ότι όχι δεν ξέρουμε ποια είναι η λύση είναι πως έχουμε αντίσταση στα κράτη-μέλη και η αντίσταση οφείλεται γιατί ακριβώς δεν θεωρούμε εαυτούς έναν ευρωπαϊκό δήμο. Είμαστε Ολλανδοί, Γερμανοί, Φιλανδοί και οι άλλοι είναι Πορτογάλοι, Ιταλοί, Έλληνες και να κοιτάξει την πάρτη τους. Αυτά και σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, σας ευχαριστώ για την τόσο ρεαλιστική ανάλυση σας. Πραγματικά. Ο ε, κύριος Ματίας Κουμ, καθηγητής, είναι αυτή τη στιγμή καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και έχει διδάξει στα πιο σημαντικά πανεπιστήμια του κόσμου και είναι και μέλος ε, της Συντακτικής Επιτροπής πολλών επιστημονικών επιθεωρήσεων και περιοδικών. Έχετε αμέσως το λόγο. Now I beg your Τώρα ζητώ την επίοικιά σα, γιατί πραγματικά καλούμε να πραγματοποιήσω μια δύνατη αποστολή. Όχι μόνο έχω 12 με 15 λεπτά για να αναπτύξω ένα περίπλοκο ε, επιχείρημα, αλλά ε, θα μιλήσω μετά τον Γιώζεφ Βάιλερ. Είναι πολύ δύσκολο να πω οτιδήποτε που δεν θα φαίνεται χλωμό και καθόλου πιστικό σε σχέση με αυτά που ακούσαμε από τον ε, καθηγητή Βάιλερ. Θα ήθελα να κάνω δύο βασικέ δηλώσει, δύο βασικέ παραδοχέ και να δώσω και κάποια επιχειρήματα. Και οι δύο παραδοχέ αυτέ δεν είναι ιδιαίτερα πρωτότυπε. Καταρχήν, η πρώτη παραδοχή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται πραγματικά δικού τη ίδιου πόρου. Και δεύτερον, οι ευρωεκλογέ θα πρέπει να μετατραπούν σε εκλογέ για να γνήσει Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και οι δύο αυτέ οι ιδέε και οι δύο αυτέ οι σκέψει ε, που θα τις βρείτε και στο έγγραφο που έχω μοιράσει και ε, περιλαμβάνεται και στο έγγραφο του κ. Μαντούρο, δεν ήταν το πρώτο. Ε, αυτό που θα ήθελα να κάνω θα ήταν να, σας παρουσιάσω ένα συγκεκριμένο επιχείρημα γιατί είναι σημαντικό να τρέξουν και τα δύο και οι δύο προϋποθέσεις και να τις ε, συνδέσω με την ε, παρούσα κατάσταση, τη συγκεκριμένη κρίση του ευρώ που αντιμετωπίζουμε. Καταρχήν, ας επικεντρωθούμε στην κρίση του ευρώ. Τι είδους κρίση είναι αυτή. Ένας λόγος είναι ότι αυτό είναι το πρόβλημα μιας νομισματικής ένωσης που δεν συνοδεύεται από δημοσιονομική ένωση. Το πρόβλημα των ασυμμετρικών συγκρούσεων, των ασυμμετρικών σοκ. Επίσης, αυτοί που σχεδίασαν τη συνθήκη του Μάστριχτ τι θα έλεγαν. Θα έλεγαν ότι εμείς δημιουργήσαμε κάποιες προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την αποτροπή αυτών των ασύμμετρικών σοκ. Βέβαια θα έσφαλα να έλεγα κάτι τέτοιο. Γιατί όμως, γιατί τα ασύμμετρικά σοκ δεν είναι, σοκ, δεν είναι σαν θεομηνίες ή μετεωρίτε που χτυπούν τη γη. Συμβαίνουν εξαιτία τη ανθρώπινη συμπεριφορά. και κάποιων αρχών που περιλαμβάνονται στις ε, στην νομοθεσία. Τι ακριβώς πήγε στραβά λοιπόν. Αυτό που πήγε στραβά, ένα από αυτά που πήγα στραβά είναι ότι κάποια, μερικά, αρκετά κράτη-μέλη τελικά ε, παραβίασαν τους κανόνες ε, διασπαθίζοντας ε, χρήματα και παραβιάζοντας τους κανόνες του Μάστριχτ για τη δημοσιονομική πειθαρχία. Οπότε ε, θα μπορούσε να πει κανείς ότι η κρίση οφείλεται στην υπερβολική σπατάλη κάποιων χωρών που, αγόρασε, που είχαν με χαμηλά επιτόκια δάνεια και μετά δημιουργήσαν ε, τεράστια χρέη και προβλήματα σε, στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης. Βέβαια υπάρχει και κάτι που αληθεύει στο στοιχείο αυτό, είναι ότι πολλές χώρες μέλη αγνώρισαν τους κανόνες σε σχέση με την ε, δημοσιονομική ευθύνη που περιλαμβάνει η συνθήκη του Μάστριχτ. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή έχουμε, 23, ε, έχουμε προσφυγές και διαδικασίες για υπερβολικό ε, έλλειμμα κατά 23 χωρών μελών. Οπότε συμβαίνει αυτό όχι μόνο γιατί ήταν σπάταλες μερικές κυβερνήσεις. Ε, συνέβη αυτό, αλλά αυτό δεν είναι ο λόγος της κρίσης. Και σίγουρα η Γαλλία και η Γερμανία, η Ιρλανδία και η Ισπανία και πολλά ε, η Γερμανία και η Γαλλία ήταν από τις χώρες που ξόδευαν περισσότερο, ενώ η Ιρλανδία και η Ισπανία θεωρούνταν από τις πιο ε, συνετές ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς αυτό. Οπότε ούτε ε, αν βρούμε ποιοι ήταν οι πιο σπάτελοι θα μας βοηθήσει να αναγνωρίσουμε τις αιτίες της κρίσης. Οπότε ποια είναι μια πιο πιστική ε, ανάλυση. Ε, ο βασικός λόγος, όχι ο μοναδικός. Αν έπρεπε όμως να επικεντρωθούμε σε ένα μόνο και λόγο για να μην δημιουργήσουμε μια πιο περίπλοκη εικόνα. Ο μόνος λόγος, αν είχαμε μόνο ένα λόγο και πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό, είναι η μεταφορά χρήματο από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα και στο χρηματοπιστωτικό τομέα ιδιαίτερο, στι Τράπεζε δηλαδή. Και εδώ ένα στοιχείο θα σα δώσω μόνο, ε, γιατί δεν προλαβαίνω μέσα στο τέταρτο που έχω. Από τον Οκτώβριο του 2008 μέχρι τον Οκτώβριο του 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε άδεια για 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ κρατικών ενισχύσεων υπέρ του χρηματοπιστωτικού κλάδου. 4,5 τρισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 33% περίπου του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Δηλαδή περίπου 6 φορές το βασικό κεφάλαιο που συνεισέφεραν τα κράτη-μέλη για τον μηχανισμό σταθερότητας. Τεράστιο ποσό. 33% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ που αναφερούνταν από, τον, από το δημόσιο χρέος, δεν θα μιλούσαμε πια για κρίση δημόσιου χρέους. Ίσως μόνο η Ελλάδα θα είχε πρόβλημα, αλλά οι υπόλοιπε χώρες δεν θα είχαν πια πρόβλημα. Οπότε στην καρδιά της κρίσης εδώ βρίσκεται μια κρίση ρύθμισης ε, του ιδιωτικού τομέα και κυρίως του χρηματοπιστωτικού τομέα των τραπεζών ώστε τα προβλήματα στον τομέα αυτό να μην μετακυλίονται στους φορολογούμενους. Τώρα, γιατί είναι σημαντικό να μιλούμε για τη Δημοσιονομική Ένωση και την σημασία που έχει να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση ίδιους πόρους. Αν πιστεύουμε, αν πιστεύετε ότι η βασική αιτία της κρίσης είναι τα προβλήματα στις, στις τράπεζες, και στη ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού κλάδου, θα μπορούσε κανεί να πει ότι ένα τμήμα της αρχική Ευθύνη ε, και τη ε, ρυθμιστική αποτυχία, ένα τμήμα της ευθύνη για τη ρυθμιστική αποτυχία θα έπρεπε να την επομιστεί από την αρχή η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή η κοινότητα των Ευρωπαίων πολιτών, αυτό ως αφετηρία. Και αυτό για πολύ απλούς λόγους, γιατί χωρίς ε, νομισματική ένωση και χωρίς ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων δεν θα είχαμε την κρίση που αντιμετωπίζουμε σήμερα με αυτή τη μορφή. Και μάλιστα όταν μια χώρα έρχεται και διασώζει τις τράπεζές της, όταν η Ισπανία δίνει 100 δισεκατομμύρια για να σώσει τις τράπεζές της, ε, αυτό ε, ουσιαστικά ε, σώζει το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αλλιώ θα είχαν τεράστια προβλήματα βασικέ τράπεζε και άλλων τραπεζών. Αυτή η ιδέα του συντονισμού τη ε, ρυθμιστική συνυπευθυνότητα μα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι από κανονιστική άποψη τέτοιες, ε, τέτοια χρέη θα έπρεπε από την αρχή να, να θεωρούνται ως πραγματικά ως γνήσια ευρωπαϊκά χρέη και να αναλυφθούν από το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια αυτό είναι ε, αυθαίρετος προς την κατανομή του κόστους ε, και της, ε, της ζημίας ανακράτος, ανάλογα με το που έχει έδρα κάθε τράπεζα. Βέβαια, θα, θα καταλήγαμε σε αυτό το συμπέρασμα μόνο αν θεωρούσαμε ότι το πρόβλημα το δημιουργεί μόνο ο τραπεζικό τομέας. Αν θεωρούμε το πρόβλημα προέρχεται από τη σπατάλη ορισμένων νοτίων χωρών, τότε θεωρούμε ότι αν οι υπεύθυνε είναι οι σπάτερε χώρε, τότε αυτέ θα πρέπει να πληρώσουν τα σπασμένα και οι επιχειρήσει του. Και μόνο ω έσχατη λύση και μόνο υπό πολύ αυστηρέ προποθέσει ε, θα μπορούσε κανεί να ασκήσει την αλληλεγγύη και να μεταφέρει χρήματα από μία χώρα σε άλλη. Αν όμω μιλούμε για μια κατάσταση όπου ήδη από την αρχή ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη κάτι τέτοιο, δηλαδή ως ένα πρόβλημα που είναι αμυγός ευρωπαϊκό, μια αμυγός ευρωπαϊκή κρίση που σχετίζεται με τους κινδύνους μιας χρηματοπιστωτικής αγοράς που εξαρτάται από τη διάρθρωση των ευρωπαϊκών κανόνων, τότε το σημείο φετηρία θα πρέπει να είναι ότι θα πρέπει να βρούμε μια συλλογική απάντηση για το χρέο ω Ευρωπαίοι. Και σε αυτό το πλαίσιο ο μηχανισμός μεταφοράς που έχουμε αυτή τη στιγμή, κυρίω μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού σταθερότητα, ε, μεταφορές δηλαδή μεταξύ των κρατών, είναι σημαντικό. και επίση θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που είπε ο κύριο Βάιλερ για την ε, Δημοσιονομική Ένωση και την έννοια του Δήμου. Θα ήθελα να σας πω μια διαφορετική ιστορία. Όχι ε, για τις συζητήσεις αν θα έπρεπε να διασωθεί η πολιτεία του Τέξας. Είναι μια ιστορία από τη Γερμανία και αφορά το Länder Finance Ausgleich. Και θα σας ε, εξηγήσω αυτή την ιστορία. Η κυβέρνηση της Γερμανίας ε, εισπράττει τους φόρους, συλλέγει τους φόρους που πηγαίνουν στην ε, ομοσπονδιακή κυβέρνηση για τις ομοσπονδιακές πολιτικές. Ένα τμήμα της όμως δίνεται στα ομόσποδα. κρατήδια. Από τα χρήματα αυτά που πηγαίνουν στα ομοσπονδιακά κρατήδια, μετά την κατανομή τους στα κρατήδια, ένα τμήμα, ένα πολύ μικρό τμήμα, ανακατανέμεται ανάλογα με τις διάφορες ανάγκες των επιμέρους κρατηδίων. Υπάρχει μια ανακατανομή λοιπόν κάποιων κονδυλίων από τα ομοσπονδιακά κονδύλια στα ομόσπονδα κρατήδια. Στη Γερμανία δεν υπάρχει καμία συζήτηση για το αν τα ομόσπονδα αν τα κονδύλια που ξοδεύονται είναι πραγματικά ομόσπονδα και πια προέρχονται από τη Βαβαρία και εξοδεύονται στη Βαβαρία, από τη στιγμή που προέρχονται από τα γενικά ομόσπονδα κονδύλια. Και το ίδιο ισχύει για τα υπόλοιπα κρατήδια. Δεν γίνονται τέτοιε συζητήσει στην Γερμανία. Όταν όμω ε, φτάνουμε στο Länder Finance Ausgleich, αυτή την ανακατανομή από το ένα ομόσπονδο κρατήδιο στο άλλο, από τη Βαυαρία στο Βερολίνο, όταν έχουμε τέτοια, τέτοιες επιμέρους μεταφορές, τότε έχουμε σφοδρή πολιτική συζήτηση και μεγάλη δυσαρέσκεια, διαμαρτυρίες και ε, δημιουργείται μείζον πολιτικό ζήτημα συνήθως με αυτές τις μεταφορές. Και γίνεται σφοδρή συζήτηση για τις επιμέρους ευθύνες των διαφόρων ομοσπονδοκρατήδιων. Βλέπετε λοιπόν τι καθορίζει τη σφοδρότητα τη συζήτηση ή το κατά πόσο θα γίνει συζήτηση. Εξαρτάται από ποιον προέρχονται τα κονδύλια και πώ μεταφέρονται. Είναι μηχανισμός που χρησιμοποιούμε που έχει αποφασιστική σημασία για το τι είδου συζητήσει θα γίνουν μετά. Γιατί η ταυτότητα ε, είναι ίδια. Είναι οι Γερμανοί ουσιαστικά που κατανέμουν τα χρήματα μεταξύ τους. Ανάλογα με το ποιο μηχανισμό επιλέγουμε, ξαφνικά δημιουργούμε ε, έλλειψη αλληλεγγύης, ε, δυσαρέσκεια, δυσανασχέτηση, ενισχύουμε κάποιες ταυτότητες ε, εις βάρος άλλων και δεν δημιουργούμε μια ευρύτερη κοινή ταυτότητα. Αν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει ίδιους πόρους και συγκεντρώσει εισπράττει χρήματα όχι από τα κράτη-μέλη, δεν θα μιλάμε για μεταφορές στην Ένωση, αλλά για τους Ευρωπαίους πολίτες ή για επιχειρήσεις ή για όποιους τέλος πάντων καταβάλουν τους φόρους και οι τράπεζες και θα μιλούσαμε για την, για την δημιουργία οικονομικής δικαιοσύνης στην Ένωση. Δεν θα θεωρούνταν ως μεταφορά από μία χώρα σε άλλη μεταφορά των χρημάτων αυτών, γιατί αυτό είναι που υπονομεύει την αλληλεγγύη και δημιουργεί δυσανασχέτηση ενισχύοντας την εθνική ταυτότητα. Ενώ αν έχουμε γενικά κριτήρια που θα θεσπίζονται από την ε, κοινοτική νομοθεσία και από τα χρήματα των κοινοτικών πολιτικών, οι συζητήσει που θα είχαμε θα ήταν διαφορετικέ και η αλληλεγγύη που θα ζητούσαμε από τους πολίτες επίσης θα ήταν διαφορετική. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Το δεύτερο αφορά το, την ανάγκη να μετατραπούν οι ευρωεκλογές σε, μία, σε εκλογές για μια ευρωπαϊκή κυβέρνηση. Θα σας πω τι κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να γίνει για κάτι τέτοιο και επίση θα, ε, πω, θα σας και θα αναφέρω και κάποια επιχειρήματα κατά της ιδέας αυτή. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει σχετικά απλά και πιστεύω ότι μπορεί να γίνει κιόλα, γιατί υπάρχουν πολλές φωνές προς αυτή την κατεύθυνση. Όλα τα μεγάλα κόμματα θα πρέπει να καθορίσουν έναν υποψήφιο, τον δικό τους υποψήφιο για πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και ε, να ε, κατέβουν όλοι αυτοί οι υποψήφοι σε μια πραγματική πανευρωπαϊκή προεκλογική εξαιρετία. Κάθε κόμμα θα προβάλλει τον δικό του υποψήφιο για, το, για τη θέση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και φυσικά θα ξέρουμε θα είναι, ποιο θα είναι το επιτελείο του, οι υπουργοί κατά κάποιο τρόπο, ε, οι υπόλοιποι επίτροποι που θα δημιουργούν ένα είδος κυβέρνησης. Η εκλογική εκστρατεία θα γίνεται ταυτόχρονα σε πολλά κράτη-μέλη, σε σχέση φυσικά με τα εθνικά κόμματα και θα παρουσιάζουν διαφορετικό πρόγραμμα με ξεχωριστές πολιτικές που θα προσωποποιούνται σε συγκεκριμένες ομάδες υποψηφίων. Με τέτοιου είδους προεκλογική εκστρατεία και τέτοια συμφωνία μεταξύ των πολιτικών κομμάτων να διεξαγάγουν πραγματικές προεκλογικές εκστρατείες μεταξύ των διαφόρων υποψηφίων των διαφόρων κομμάτων, πιστεύω ότι κατά πάσα πιθανότητα θα καταλήξουμε σε πολύ διαφορετική ανταπόκριση του εκλογικού σώματος και πολύ μεγαλύτερη προσέλευση στις ευρωεκλογέ, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι τώρα. Και γιατί είναι σημαντικό κάτι τέτοιο. Κάτι που φάνηκε πολύ πιο έντονα στην κρίση του ευρώ είναι ότι ένα από τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά τη γνώμη των πολιτών της, είναι ότι φαίνεται ε, ως ε, ένα μονολυθικό μπλοκ ε, αποτελεσμάτων. Αν σας αρέσουν τα αποτελέσματα, σας αρέσει και η Ευρώπη. Αν δεν σας αρέσουν τα αποτελέσματα, κατά πάσα πιθανότητα θέλετε λιγότερη Ευρώπη, θα είστε κατά της Ευρώπης. Αν σας αρέσουν τα επιτέγματα της Ευρώπης, θα θέλετε περισσότερη Ευρώπη. Ως πάντως θεσμικό μηχανισμό δεν έχουμε εναλλακτικές Ευρώπες που να παρουσιάζονται σε μια δημόσια συζήτηση για να μπορούν να πούν οι πολίτες όχι αυτή η Ευρώπη δεν μας αρέσει αλλά η άλλη Ευρώπη ίσως θα μπορούσε να μας ικανοποιήσει, θα μπορούσαμε να ταυτιστούμε με αυτή. Να υπάρχουν δηλαδή επιλογές μεταξύ διαφόρων προσανατολισμών για τους πολίτες. Αυτό υπό το πρίσμα των πολιτών θα ήταν ένα πολύ καλό αντίβαρο απέναντι σε ένα συγκεκριμένο ευρωσκεπτικισμό και ένα συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη έξαρση του εθνικισμού. Δηλαδή, η σημερινή ιδέα είναι ότι δεν σας αρέσει η ιδέα η σημερινή Ευρώπη, αλλά δεν υπάρχει καμία εναλλακτική λύση. Θα ήταν σημαντική λύση λοιπόν να δοθούν και εναλλακτικέ λύσει για την Ευρώπη. Πιστεύω ότι πολλά θα κερδίζαμε αν βαδίζαμε προ αυτή την κατεύθυνση. Το θέμα είναι, είναι ρεαλιστική αυτή η κατεύθυνση και ποιο θα είναι το τίμημα μια τέτοια απορίας. Μήπως είναι υπέρογκο. Αυτή η συζήτηση έγινε αρκετές φορές. Εγώ θα ήθελα να σας παραθέσω κάποια επιχειρήματα κατά της ε, κατεύθυνσης αυτής. Ένα βασικό επιχείρημα είναι, κοιτάξτε πώς γίνονται τώρα οι ευρωεκλογέ. Μας έδωσε κάποια στατιστικά στοιχεία ο Τζοζεφ Βάιλερ που μας δείχνουν ότι οι πολίτες ε, δεν ενδιαφέρονται περισσότερο παρά την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουμε μεγάλο ποσοστό αποχής, πολύ χαμηλότερη προσέλευση στις ευρωεκλογές από τις εθνικές εκλογές. Οπότε πρέπει να υπάρχει ένα βαθύ συστημικό πρόβλημα που δεν μπορούμε εύκολα να το υπερκεράσουμε. Και άλλοι μιλούν είτε για χαμένη ταυτότητα ή ταυτότητα που λείπει τέλο πάντων, είτε ε, ε, ένα πρόβλημα στον κοινωνικό ιστό, ίσως στην διάρθρωση των πολιτικών κομμάτων, γιατί δεν υπάρχουν ενοποιημένα πολιτικά κόνημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν υπάρχουν πραγματικά κόμματα που να ενδιαφέρονται να κρατήσουν ε, συμμαχίες μεταξύ τους. Υπάρχουν λοιπόν τέτοια προβλήματα και δεν είναι καθόλου περίεργο που βλέπουμε τι μορφή έχουν τα θεσμικά όργανα και πόσο δύσκολο είναι να αλλάξουν. Θα δούμε όμως αν κάτι τέτοιο ισχύει. Αυτό θα φανεί αν στις επόμενες ευρωεκλογέ έχουμε μια εκλογική διαδικασία πολύ πιο ανταγωνιστική από αυτή που σας ανέφερα. Πιστεύω ότι μπορούμε να τη δοκιμάσουμε, γιατί αν τη δοκιμάσουμε και γίνει σωστά και σοβαρά, πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα είναι εντυπωσιακά και η προσέλευση πολύ πιο μεγάλη. Και θα ήταν χρήσιμο να δοκιμάσουμε μια τέτοια πιο ανταγωνιστική προεκλογική εκστρατεία. Ένα άλλο αντεπιχείρημα είναι πιο ακαδημαϊκό βέβαια, αλλά υπάρχει και μια πολιτική του πτυχή και δεν θα πρέπει να την αμελήσουμε. Υπάρχει ιδέα ότι υπάρχει, υπάρχει κάτι προβληματικό και κάτι ανεπιθύμητο στην δημιουργία κάποιων χαρακτηριστικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τα, σχετίζουν, τα συσχετίζουμε με το κράτος, στην βαρετή κλασική μορφή του κράτους. Είναι έτοιμη η Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεπεράσει αυτή την κατάσταση και να δημιουργήσει κάτι αυθεντικά καινούριο. Και τώρα όσο προχωρεί η κατάσταση καταλήγουμε σε κάποια χαρακτηριστικά διαρθρωτικά που φαίνεται ότι την προσωμιάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση όλο και περισσότερο με ένα κλασικό κράτος. Τέτοιο τους επιχείρημα θα μπορούσε να καταρριφθεί με, ε, με την ευαισθησία, η παρόμοια ευαισθησία με αυτή που έδειξε ο Ζαμονέ καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Εκείνος δεν ενδιαφερόταν για τις περιγραφές, αν την πρότασή του τη χαρακτηρίζεται διεθνή οργανισμό ή ιδιότυπη οντότητα, σου generis οντότητα. Αυτό που ενδιαφέρει τον Σάμονε είναι να υπάρχουν ε, λειτουργικοί αποχρόντες λόγοι για να συγκεντρωθούν οι πόροι και για κοινή συνεργασία. Και η, ιδέα του, η βασική, είναι ότι υπάρχουν κάποιες θεμελιώδεις ε, αξίες πίσω από την ιδέα αυτή. Και αν ε, καταλήξουμε ότι είναι σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει κάποιε αρμοδιότητε και στο δημοσιονομικό τομέα. Και αν καταλήξουμε ότι υπάρχουν αποχρόντε λόγοι για να δημιουργηθούν μηχανισμοί ε, εκλογική ε, λογοδοσία κάτι σαν κυβέρνηση και πραγματική πολιτική, γνήσια πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τότε αν είμαστε πεπισμένοι γι' αυτό θα πρέπει να το κάνουμε και να μην ε, μας εκφοβήσουν αυτοί που χρησιμοποιούν τον όρο υπερκράτος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να εμείνουμε σε έναν ρεαλισμό, ε, σε μια σταδιακή πορεία λειτουργική όπως αυτή που ακολούθησε ο Ζαν παρόλο που διανύουμε χαλεπούς καιρούς ε, γιατί ε, παρόλο που μπορεί κάποια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει δομές παρόμοιες με αυτές που μας είναι οικίες από τα έθνη κράτη. Ευχαριστώ. <clears throat> Ευχαριστώ καθηγητά κύριε Κουμ. Και τώρα θα δώσουμε το λόγο στον καθηγητή κύριο Μαντζέλα ο οποίος διδάσκει κοινοβουλευτικό δίκαιο στο Πανεπιστήμιο Λούι στη Ρώμη, πρώην δικαστής και πρώην ευρωβουλευτής από το 1994 στο 1999. Παρακαλώ, έχετε το λόγο κύριε Μαντζέλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα μιλήσω Ιταλικά. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ε, βάλτε τα ακουστικά σας. Θα ε, ήθελα στο μεταξύ να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση αυτή. Ε, με τιμά και με γυρίζει και πίσω σε ένα παλιό μου έρωτα. Ε, ε, μου τέθη ένα ερώτημα. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι νομιμοποιημένο πιευτικό θεσμικό όργανο σε μια νέα πολυεπίπεδη οικονομική διακυβέρνηση ε, στην Ευρώπη. Μάλλον πρέπει να το αντιστρέψουμε το ερώτημα και να αναρωτηθούμε περισσότερο εάν η νέα οικονομική διακυβέρνηση ε, χαρακτηρίζεται από μία νομιμότητα ίδια και σε ποιο βαθμό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, βοηθάει στην επίτευξη αυτής της νομιμότητας. Ποια είναι τώρα η καινοτομία ε, στη συζήτηση. Ε, το θέμα του δημοκρατικού ελλείμματος άλλαξε φύση. Πριν τη μεγάλη κρίση αυτό φαινόταν ε, να αφορά μόνο τις μεγάλες σφαίρες και τους υψηλούς κλάδους των τεσσάρων θεσμικών οργάνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφενός και την ε, Ευρωπαϊκή Κοινή Γνώμη, το λαό από την άλλη ή τον Ευρωπαϊκό Δήμο ανάλογα με τις διάφορες ερμηνείες. Τώρα, το θέμα του δημοκρατικού ελλείμματος ή μάλλον της ε, νομιμότητας έχει ε, καταστεί αδιέρετο, δηλαδή αφορά ε, πλέον το στο σύνολό της και την Ένωση αλλά και τα κράτη, γιατί έχουν μία κοινή πολιτική μοίρα. Δηλαδή, η κρίση της δημοκρατικής πράξης περιέργως και παραδόξως έχει οδηγήσει ε, με αρνητικό τρόπο σε ένα βαθμό ολοκλήρωσης της Ένωσης και των κρατών μεταξύ τους που κανένα θετικό μέτρο μέχρι τώρα δεν είχε καταφέρει να επιτύχει. Τι συνέβη στην Ένωση με τη μεγάλη κρίση οι εθνικές ε, δυναμικές συμπιέζονται και οι εξουσίες των κυβερνήσεων αλλά ακόμα και οι εξουσίες των κοινοβουλίων στην επικράτειά τους. Το πρόγραμμα των δημοσίων πολιτικών πλέον έχει ένα ετερόφωτο χαρακτήρα, δηλαδή ε, έξωθεν ε, αποδίδεται αυτό και ισχύει κυρίως για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και ε, νομικά αυτό επισημοποιείται στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Δηλαδή, ποντάρουμε πλέον σε ένα φεντεραλισμό και σε ένα κοινοβουλευτισμό εκτελεστικής φύσεως. Έχουν αρχίσει να διαβρώνονται ίσως οι συνθήκες. Ποιος είναι κυρίαρχος. Κυρίαρχος των συνθήκων είναι τα κράτη, αλλά ε, πλέον από κοινού. Ε στο βαθμό που όλοι μαζί συμφωνούν το κοινό πλαίσιο. Ο βασικός μηχανισμός λοιπόν των κοινωνικών καθεστώτων έχει αλλάξει. Ε, Δηλαδή, ε, έχει διπλασιαστεί. Οι κυβερνήσεις δεν χρειάζονται μόνο την πίστη των κοινοβουλίων τους, αλλά και την πίστη των θεσμικών οργάνων. Και ο μηχανισμός ε, της κοινοβουλευτική μορφή, η δυσπιστία δηλαδή και παρέτησης, ε, υπολείπεται κατά πολύ σε σχέση με μια ευρωπαϊκή δυσπιστία ως προς την κύρωση, γιατί υπάρχει κύρωση της αντίδρασης των αγορών, που είναι πραγματικά ένας βραχίωνας πλέον επιβολής ε, ε, οικονομικών υποχρεώσεων. Έτσι λοιπόν η μεγάλη κρίση έχει καθορίσει αυτό το πλαίσιο, αλλά και σε κρίσιμες συνθήκες αυτό που ε, πάντα ονειρεύονταν οι ευρωπαϊστές και ο Βάιλερ. Δηλαδή, τι ονειρεύονταν. Τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δημοσίου χώρου που να χαρακτηρίζεται από το κέντρο του ευρωπαϊκού ζητήματος, το οποίο κυριαρχεί στη δημόσια συζήτηση. Ναι, αλλά τώρα έχει εκρηκτικό χαρακτήρα γιατί ε, πυροδοτεί ε, αλυσιδωτές αντιδράσεις της κυβερνήσεις ή κυβερνήσεις τεχνοκρατών ή επιτροπίες ή κυδαιμονίες ή πρόθεση ακόμα και αντιευρωπαϊκών κινημάτων ή ακόμα και κινήματα που διεκδικούν ποσοστώσεις ε, εθνικής κυριαρχίας που έχουν χαθεί. Και περιέργως οι ε, ευρωπαϊκοί θεσμοί, ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα αποφασίζουν και ακολουθούν οι εθνικοί θεσμοί. Όχι σαν πυροσβέστες οι οποίοι έρχονται να ε, ε, συγκρατήσουν μια πυρκαγιά, αλλά πυρομανείς οι οποίοι πυροδοτούν τις καταστάσεις. Έχει αρχίσει λοιπόν και γεννιέται μια ιδέα ευρωπαϊκού, πανευρωπαϊκού δημοψηφίσματος. Δηλαδή μέσω της άμεσης προσφυγής στο λαό και οι κυβερνήσεις και οι δικαστές, οι εθνικοί και τα κοινοβούλια ε, ε, προσπαθούν να αποποιηθούν των ευθυνών τους γιατί η κοινή γνώμη είναι όλο και πιο ε, επιθετική και όλο και πιο ανήσυχη. Απέναντι λοιπόν σε αυτές ε, τις καταστάσεις και τους κινδύνους για την Ένωση και για τα κράτη-μέλη, ο ρόλος του Κοινοβουλίου δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στην μία ή στην άλλη του ιδιότητα ή αποστολή. Θα πρέπει να δραστηριοποιείται ε, αλλά σε ποιο επίπεδο, στο κοινοτικό, στο εθνικό, θα πρέπει να υπάρχει ένα κύκλωμα ε, δημοκρατικής νομιμότητας που να είναι πιστική στα μάτια της κοινή γνώμης. Θα έλεγα λοιπόν, και αυτό θα λέει και ο καθηγητής Ντεούς, εδώ έρχεται ο ερμηνευτής να ε, αξιολογήσει τι γίνεται με την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση και ποιο είναι το δυναμικό που φέρνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να υπάρξει ε, μια πρόοδος δημοκρατική συλλογική. Τι βλέπουμε το τελευταίο διάστημα. Τρεις αλλαγές σε βάθος. Πρώτη αλλαγή. Η προσφυγή στο διεθνές δίκαιο για να ξεπεραστεί η εμπλοκή ε, που ε, υφίστανται ορισμένα κράτη για να λάβουν νέα μέτρα δημοσιονομικής σταθεροποίησης. Το δεύτερο είναι η εισβολή ε, στο συνταγματικό δίκαιο των κρατών μελών για να υπάρξει ε, ομοιογένεια δημοσιονομική και τρίτον, ε, πώς να το πω, πώς να το χαρακτηρίσω, υπάρχει μια νέα εφεύρεση εφεύρεση είναι αυτή ε, διακοινοβουλευτικής συνεργασίας μονίμου χαρακτήρα, διαρκής είναι αυτή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις εθνικές Βουλές. Σε ό,τι αφορά το πρώτο, το διεθνές δίκαιο, φαίνεται προφανές ότι το δημοσιονομικό σύμφωνο και το σύμφωνο για τη, του σταθεροπικού μηχανισμού που είναι μια δορυφορική συνθήκη, γιατί υπάρχει και αυτή η ρήτρα, ε, πώς τη λένε, χρησικτησίας, περιπτώσει, ε, ε, αυτή τη στιγμή ε, εγκριθεί και κυρωθεί. Σε ό,τι αφορά αυτό το πρώτο λοιπόν για το Δημοσιονομικό Σύμφωνο, θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει μια ενισχυμένη συνεργασία με άλλα μέσα για να ξεπεράσει τα τυπικά εμπόδια που είπε ο κύριος Ντεβίτ ότι υπάρχουν τυπικά εμπόδια ε, και τα πολιτικά εμπόδια για τη ε, χρηματοοικονομική σταθεροποίηση. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως προβλέπονται στις συνθήκες της Αβώνας διατηρούνται στο ακέραιο σε κάθε πτυχή τους, αλλά ενισχύονται εάν αξιολογούμε και τις σχέσεις που έχει με τις νέες ε, λειτουργίες ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή, έχει το συνήθι κοινοβουλευτικό έλεγχο το κοινοβούλιο. Αλλά ε, υπάρχει και μία νέα αποστολή ε, συμμετοχής και ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα πρέπει να το δούμε από δύο σημεία. Πρώτον, σε αυτή την άτυπη ενισχυμένη συνεργασία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην ολομέλεια του και με τον αδιέρετο χαρακτήρα του έχει ένα δικαίωμα ε, λόγου ε, παρόλο που ευρωβουλευτές ε, εκλέγονται σε χώρες εκτός αυτής της συνθήκης του Δημοσιονομικού Συμφώνου δηλαδή. Στο δεύτερο σημείο Ε, επίσης, ε, πάλι έχει ένα διέρατο χαρακτήρα, γιατί οι ευρωβουλευτέ προέρχονται από χώρες της Ευρωζώνης και χώρες εκτός της Ευρωζώνης. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται να συζητήσει, ε, όπως λέει το άρθρο 13 του Δημοσιονομικού Συμφώνου, τις ε, πολιτικές με τις αρμόδιες ε, ομόλογες επιτροπές των Εθνικών Κοινοβουλίων. Δηλαδή, σε αυτά τα δύο σημεία που καταρχήν επιβεβαιώνουν την αρχή του αδιαιρέτου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, απορρίπτεται η ιδέα λοιπόν ενός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με μεταβλητή γεωμετρία. Αν σκεφτούμε πώς έχει σήμερα το πανόραμα ε, και η μεγαλύτερη ε, διαφοροποίηση στην Ευρώπη, η ενότητα του Κοινοβουλίου είναι από μόνη της ε, ένας παράγων δημοκρατικής νομιμότητας. μάλιστα θα χαρακτήριζα ένα μπλοκ νομιμότητας απέναντι στην μεταδοτικότητα του διεθνισμού και του διακυβερνητισμού. Για το δεύτερο, εισβολή ε, στην ένωμη τάξη, στην ταγματική των κρατών μελών. Είτε πρόκειται για το ευρωπαϊκό εξάμεινο ή την υποχρέωση ισοσκελισμένου προπολογισμού ή ακόμα και το δημοσιονομικό σύμφωνο ε, να τίθεται σε ισχύ ε, εγκαταλείποντας την αρχή της ομοφωνίας. Δηλαδή συνδέεται η βοήθεια του μηχανισμού σταθερότητας με την έγκριση του Δημοσιονομικού Συμφώνου. Εδώ λοιπόν έχει ρόλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, στη χάραξη των νέων κανόνων με τους ΣΕΡΠΑ που συνεδριάζουν, ε, ξέρετε, σαν να είχαν ήδη προβλέψει τη μέθοδο των διαβουλεύσεων ε, της ε, δήλωσης παριθμών 11. Είναι γεγονός ότι αυτή η σημαντική παρουσία δεν αντανακλάται στις αρμοδιότητες και τις λειτουργίες που παραχωρούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα. Σαν να ήταν σήμερα ένα όργανο που ε, ενδιαφέρεται μόνο για τη συντάγμα γενικά, αλλά δεν συμμετέχει στους άλλους μηχανισμούς. Ε, είναι όμως πολύ σημαντικός ο οικονομικός διάλογος και συμμετείχε το Κοινοβούλιο με το εξαπλό πακέτο, θυμάστε το πακέτο των έξι οδηγιών. Και επίσης ο διάλογος που μπορεί να βαρύνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την πλειοψηφία του, αλλά και από το γεγονός ότι είναι και σκέλος της δημοσιονομικής αρχής με όσα ε, συμπαραμαρτούν τα προβλήματα γνωρίζουμε και έχουμε δει. Αλλά και ο προϋπολογισμός είναι η καρδιά ε, και πάντα της δημοκρατικής διαβίωσης. Το τελευταίο, τρίτο στοιχείο. Η σχέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Δίνεται η εντύπωση ενός άλματος προς τα εμπρό σε σχέση με τη Λισαβόνα. Αλλά, ε, και βεβαίως σε συνοχή με και συνάφεια με τη Λισαβόνα, αλλά... Υπάρχει και κάτι ακόμα. η ιδέα ενό γνήσιου ευρωπαϊκού κοινοβουλευτικού συστήματο με αυξημένο ρόλο για τα εθνικά κοινοβούλια και ιδιαίτερα διακοινοβουλευτική συνεργασία. Πώς να το πω. Σε αυτή τη διακοινοβουλευτική συνεργασία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί ε, ε, ρεαλιστικά να έχει ένα ρόλο κλειδί. Είναι εκείνο που θα έχει ε, το κλειδί για, για τις διάφορες ε, διασκέψεις και το δίκτυο. Δηλαδή είναι ένας κοινοβουλευτισμός διασύνδεσης, να το χαρακτηρίζα. Ε, ψηφίζουν τα εθνικά κοινοβούλια, αλλά δεσμεύονται και από την ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βεβαίως, σήμερα Ξέρουμε ότι υπάρχουν αντιρρήσεις απέναντι σε ένα κοινοβούλιο που θα εκπροσωπεί τα κράτη, μέλη, σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά ε, θα πρέπει να είναι μια ένα σώμα διαβούλευσης ε, και πέρα από το σώμα ε, διαβούλευσης αμυγός ή απόφασης υπάρχει και ένα ενδιάμεσο σώμα, ένα σώμα άσκησης επιρροής και ακόμα και νομικά ισχύει αυτό το επιχείρημα ε, σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο. Συνοψίζω, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε πραγματικά να διαδραματίσει ένα ρόλο ε, δικτύωσης με κοινοβουλευτικές διασκέψεις και να διατηρείται έτσι ώστε να υπάρχει γνήσια και πραγματική ε, ε, ουσία στη διακοινοβουλευτική συνεργασία. Σύνοψίζοντα ε, Πρόεδρε, και καταλήγοντα, θα έλεγα ότι οι νέε διαστάσει τη οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρώπη δεν ε, μειώνουν, δεν είναι επιβλαβής για τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αλλά χρειάζεται και μια κάθετη δομή πέρα από την εγκάρσια. Όταν γίνεται λόγος για την ομιμοποίηση του Κοινοβουλίου, Βεβαίως το Κοινοβούλιο έχει ενεργό ρόλο ως νομοθέτης, αλλά χρειάζεται και μια άλλη νομιμοποίηση, η οποία μπορεί να έλθει μόνο ε, από την ποιοτική ε, ψήφο του λαού και των πολιτών. Και ε, ένας εξωτερικός παρατηρητής απορεί για τις απόπειρες που έχουν αβαγίσει μέχρι τώρα, όπως του κυρίου Νταφ και άλλων, ε, το είπε και ο καθηγητής Κουμ, δηλαδή η ιδέα ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα μπορούν να κάνουν πολλά, οι ευρωπαϊκές πολιτικές παρατάξεις, για να αποεθνικοποιήσουν την ψήφο στις ευρωεκλογές των Ευρωπαίων πολιτών για να είναι γνήσιες ευρωπαϊκές οι ευρωεκλογές, οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μέχρι το 2014 υπάρχει ακόμα χρόνος για να εργαστούμε. Βέβαια δεν είναι απεριόριστος και ανεξάντλητος, αλλά υπάρχει χρόνος και θα πρέπει να αξιοποιηθεί. Διότι είναι ψευδέστηση να πιστεύει κανείς ότι η νομιμοποίηση μπορεί να έλθει μόνο ε, από την εξάπλωση, το spillover των οικονομικών ε, μέσων, όσο καινοτόμα και να είναι αυτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Μαντζέλα. Κλείνει εδώ η δεύτερη σύνοδος. Ποια είναι η δεύτερη, η τρίτη σύνοδος του σημερινού σεμιναρίου. Ακούσαμε ε, τους ε, πέντε ομιλητές ε, και θα μιλήσουν οι συνάδελφοι. Πρώτος ο συνάδελφος Τσαρκόφσκι. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τις τρεις εξαιρετικέ αυτές παρεμβάσεις. Τι θέλω να κάνω. Θέλω πρώτα να κάνω δύο σχολεία και μετά μια ερώτηση. Αναφερθήκατε σε πολλά ζητήματα. Τώρα ξεκινώντας με αυτό το οποίο είπε ο κύριος Βάιλερ για την αλληλεγγύη και τον Δήμο γιατί κάνατε αυτή τη σύγκριση με το Τέξας και την Καλιφόρνια ή τη Μασαχουσέτη και ξέρω εγώ τι ε, εσείς πάντα γράφατε για τον Δήμο και ότι κάνουμε τη συνειδητή επιλογή να μην δημιουργήσουμε ένα Δήμο και ότι δεν θα πρέπει να έχουμε αυτό το στόχο. Αναρωτιέμαι εάν αυτό είναι πραγματικά ζήτημα ύπαρξη Δήμου ή όχι. Γιατί για να πάει κανείς και στην ιστορία των ΗΠΑ τη συζήτηση μεταξύ Μάντισον και Χάμιλτον για την ε, δημοσιονομική ευθύνη ήταν ακριβώς η ίδια με αυτή την οποία έχουμε τώρα και τα επιχειρήματά τους ήταν τα ίδια. ω κάποιες πολιτείες η, πολι... Βιργίνια πλήρωνε το χρέο τη και οι υπόλοιποι τη βγάζανε τζάμπα εις βάρος των υπευθύνων και αυτό είχε βεβαίως την ε, πιθανότητα να, να γυρίσει μπούμεραγκ. Τόσο δεν θα ξεκινήσουμε τώρα τη συζήτηση για το αν υπήρχε Αμερικανικός Δήμος τότε, αλλά υπήρχε οπωσδήποτε τότε πολύ περισσότερος από όσο θα έχουμε εμείς ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αντιλαμβάνουμε και τη γερμανική συζήτηση όταν λένε ότι ναι, το να δώσουμε λεφτά στους Πολωνούς με τα διαρθρωτικά κονδύλια και να τα χρησιμοποιούν σωστά, εντάξει δεν είναι πρόβλημα γιατί συμπεριφέρονται υπεύθυνα και βλέπω πού πάνε τα λεφτά μου, δηλαδή πάνε για ένα καλό σκοπό. Ενώ το να δώσουμε λεφτά στους Έλληνες, όχι, γιατί δεν είναι υπεύθυνοι. Αυτό υπάρχει στη γερμανική δημόσια συζήτηση. Το είχε πει ο Σόιμπλε, νομίζω, υπουργό Οικονομικών. Και πολλοί Γερμανοί συμφωνούν μαζί τους. Ότι δηλαδή, εντάξει, να δίνουμε λεφτά στους υπεύθυνου, το καταλαβαίνω. Είναι μια ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και παράγει και δουλειέ στη Γερμανία κτλ. κτλ. λοιπόν, εάν είναι ζήτημα ε, μιας κοινή μοίρα ή όχι, αντί για ζήτημα Δήμου. Επίσης ε, το θέμα Και επίσης ε, για το θέμα που αναφέρατε, το αν μπορούμε να διώξουμε τα, καθάρματα, εάν είναι αυτό ένα πραγματικό πρόβλημα. Ε, δηλαδή, πέραν του, αποκεφαλισμού του Προέδρου της Κομισιόν ε, όταν τελειώσει η θητεία του και δεν αρέσουν τα αποτελέσματά του, δεν ξέρω ποια λύση θα μπορούσαμε να έχουμε για να συγκλονίσει τον κόσμο. Δηλαδή, στην Επιτροπή μας, ναι, εμείς είμαστε υπέρ του να έχουμε, παραδείγματος χάρη, ε, Ευρωεκλογέ ε, με πολιτικά κόμματα και να λέει το ΕΛΚ αυτόν έχουμε εμεί υποψήφιο για πρόεδρο, αυτό είναι το πρόγραμμά μας και να κάνει μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία κάτω από αυτό το, το λάβαρο. Ναι, μια πολύ καλή ιδέα και εμεί υποστηρίζαμε κάποιοι τουλάχιστον την ιδέα του να έχουμε μια υπερεθνική λίστα τουλάχιστον για ένα μικρό αριθμό βουλευτών κάτι το οποίο βεβαίως απέριψε η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου και, και αυτό σας λέει κάτι αλλά δεν είμαι σίγουρος, παρά το ότι ευχαρίστως να, να ξεκινήσουμε αυτό το πείραμα, δεν είμαι σίγουρος ότι θα άλλαζε τίποτα. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Το πρόβλημα είναι πως ο κόσμος θεωρεί πως το ευρωπαϊκό επίπεδο δεν μου λύνει τα προβλήματά μου. Τα προβλήματά μου είναι απασχόληση, εκπαίδευση, υγεία, συντάξεις. όλα αυτά είναι στο εθνικό επίπεδο. Ανεξάρτητος το αν έχουν δίκιο ή όχι. Και ακόμα και αν δίναμε αυτή τη δυνατότητα κάποια επιρροή στην κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα άλλαζε τίποτα. Επιπλέον αυτό υπάρχει ε, εγγενές στο πολιτικό μας σύστημα. Δηλαδή διαφέρουμε τόσο πολύ, ε, εγώ είμαι από το ΕΛΚ κεντροδεξιά, διαφέρουμε τόσο πολύ από τους σοσιαλιστές όταν μιλάμε για τις απόψεις μας για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, εντάξει, προφανώς υπάρχουν κάποιες διαφορές, αλλά είναι αρκετά μεγάλες. Εδώ μέσα παραδείγματο χάρη υπάρχει μια κουλτούρα συμβιβασμού, εγγενής στο σύστημα. Εντάξει, τσακωνόμαστε, διαφωνούμε, αλλά σε τελική ανάλυση καθόμαστε, εμείς δηλαδή, οι σοσιαλιστές, φιλελεύθεροι και ΕΛΚ και συμβιβαζόμαστε γιατί αλλιώς δεν θα καταφέρουμε τίποτα σε σχέση με τα κράτη-μέλη και τις διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο. Και ποτέ δεν θα υπάρξει εδώ μέσα πλειοψηφία, μειοψηφία δηλαδή. Οπότε α, οι διαφορές ε, χάνονται κάπου μέσα σε αυτή την κουλτούρα του συμβασμού και είναι δύσκολο να έχουμε τελείως διαφορετικές απόψεις. Δείτε και την Επιτροπή μας εδώ μέσα, τα μεγάλα πολιτικά κόμματα εδώ μέσα, παρά το ότι έχουμε κάποιες διαφορές, συμφωνούμε στο 95% των περιπτώσεων. Και τέλος, ένα άλλο ερώτημα. Είμαστε σε, σε μια κρίση και ο κόσμος αναζητά ριζοσπαστικές λύσεις. Κάποιοι θα πήγαιναν προς μια ομοσπονδιακή κατεύθυνση και θα έλεγαν αυτή είναι η λύση που πρέπει να εκτίσουμε, άλλοι θα ήταν σκληροί, ας πούμε, έτσι. Ο Ζαν στην πρώτη του προσέγγιση, στο βιβλίο του, ε, είχε πει πως πρέπει να δημιουργήσουμε μια ένωση με στην ένωση, με νέα θεσμικά όργανα κτλ. Αλλά εγώ πιστεύω και πάντα μας λέγατε εσείς πως πρέπει να προσπαθήσουμε να είναι πάντα μοναδικό και ενιαίο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, μια συνταγματική ανοχή κτλ. Μπορούμε ακόμα να, να κάνουμε κάτι τέτοιο. Κάποιοι λένε πως είναι το ζήτημα της διεύρυνσης, έχουμε γίνει πολύ ανομοιογενείς, έχουμε φτάσει στο σημείο που πλέον δεν είναι δυνατόν, γι' αυτό αναζητάνε αυτές τις ριζοσπαστικές λύσεις. Το ερώτημά μου είναι μπορούμε να υπερασπίσουμε το, α, το μοναδικό και το ενιαίο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, γιατί νομίζω πως αυτό είναι τελικά το ζήτημα που πρέπει να απασχολεί στην Επιτροπή μας. Ε, Andrew, the floor yours. Yes, um... Andrew. Ευχαριστώ. Ράφα που εκεί που δεν λειτουργεί συμβαστική ε, η επιθυμία συμβασμού και το πνεύμα ε, συμβιβασμού είναι στα θέματα τα φεντεραλιστικά. Οι διαφορές δεν είναι μεταξύ των κλασικών πολιτικών οικογενειών, αλλά περισσότερο μεταξύ των αυτών που είναι φεντεραλιστές και αυτών που είναι ε, εθνικιστές περισσότερο. Και ε, εγώ ζηλεύω την αμερικανική εμπειρία, γιατί τότε η δημιουργία των δύο βασικών στρατοπέδων του Κογκρέσου, των φεντεραλιστών και των ρεπουμπλικάνων δηλαδή, θυμόμαστε άλλωστε ότι ο George Washington ήταν κατά της ε, δημιουργίας ε, τότε, της ενίσχυσης εκείνης της ε, πλευράς τότε, αλλά συνέβη σχετικά γρήγορα. Δεν υπήρχε όμως ανταγωνιστικότητα μεταξύ των δύο βασικών κομμάτων στις 13 πολιτείες και εμείς αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα αλλά σε πολύ πιο περίπλοκες συνθήκες. Γιατί εκεί έχουμε άμεσο ανταγωνισμό και μάλιστα σύγκρουση με εθνικά κόμματα, εθνικά πολιτικά κόμματα και με τα δικά του συμφέροντα και μάλιστα τα εθνικά πολιτικά κόμματα έχουν μια πολύ ε, πιο κοντόφθαλμη προσέγγιση, με ένα πολύ πιο κοντόφθελο όραμα και προσβλέπουν σε, μια, σε ένα μονοπόλιο της εξουσίας. Και αυτόν που στέλνουν και εδώ και αυτόν που στέλνουν και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περιμένω με ανυπομονησία τα σχόλια και τις συμβουλές των Αμερικανών ε, συναδέλφων. Πώς λοιπόν θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ε, πανευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Και λοιπόν ειλικρινά που οι προτάσει μου για, τις, για τους πανευρωπαϊκούς εκλογικούς και τα πανευρωπαϊκά ψηφοδέλτια ε, δυστυχώς ε, δεν ευωδόθηκαν και έμειναν κάπου παγωμένες εδώ στο Κοινοβούλιο. Δεν μπορούμε βέβαια να υποχρεώσουμε τα πολιτικά κόμματα να υποβάλουν τους υποψηφίους τους, τους πρωταθλητές τους και να τους υποβάλουν στους υποψηφίους ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι σημαντικό όμως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αντιληφθεί ότι θα αναλάβει ευθύνες για την εκλογή του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάτι που δεν ίσχυε πριν τη συνθήκη της Λισαβόνας. Και από τη στιγμή που ο κύριος Μπαρόζο δεν θα ξανά είναι μάλλον υποψήφιος, ίσως πραγματικά γίνει επικρατήσει μεγάλη αντιπαράθεση για τη διαδοχή του και η τελική απόφαση θα είναι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ελπίζω πάντως ότι θα συμφωνήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να επιμείνουμε η μισή επίτροπη το 2014 να προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κάτι τέτοιο θα συμβόλιζε το χαρακτήρα που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως συνομοθέτης μαζί με το Συμβούλιο και μάλιστα έχουμε ήδη ένα προηγούμενο με τον Μισελ Μπαρνιέ που το 2009 πρώτα εξελέγει Ευρωβουλευτής και μετά μεταγράφει και μετατέθηκε, αποσπάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή λίγες εβδομάδες αργότερα μετά την εκλογή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χρειαζόμαστε λοιπόν και αυτοπεποίθηση και κάποια διορατικότητα για να κάνουμε αυτούς τους πειραματισμούς και να αναζωογονήσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχει ε, πολλούς φεντεραλιστές και ελπίζουμε να είναι πολύ περισσότεροι μέχρι το 2014. Επίσης, η διατάξει της Λισαβόνας για, τις, ε, για το μέγεθος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να τηρηθούν. Δηλαδή θέλουμε 19 επιτρόπους και όχι 28 στην Επιτροπή του 2014. Και όταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, έκανε ένα είδος χατηριού προς την Ιρλανδία για να την πείσει να δεχθεί τη συνθήκη της Λισαβόνας, ελπίζω τέτοιες χειρονομίες να μην συνεχιστούν και στην επιλογή τη, της νέας σύνθεσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και μια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πια λόγο στην έγκριση των επιτρόπων, θα έχουμε πολύ πιο καλύτερη θέση για να επιβάλλουμε αυτή την ανάγκη να τηρηθούν οι διατάξει τη συνθήκη Λισαβόνα για, για το έβρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, κύριο Μπρόν. Ευχαριστώ. Η τοποθέτηση του καθηγητή Βάιλερ νομίζω ήταν ενδιαφέρουσα και, και ειλικρινής θα έλεγα. Η δική μου η προοπτική είναι βεβαίως ξεκάθαρα εθνικιστική, αλλά δεν σημαίνει αυτό πως είμαι αδιάφορος για τα όσα υποφέρουν λαοί σε άλλες χώρες. Είναι εύκολο να περιγράψουμε την προθυμία των ευρωπαϊκών χωρών να διασώσουν τον Νότο ως κακία, η έλλειψη γενεοδορίας. Αλλά η απουσία Ευρωπαϊκού Δήμου είναι γεγονός που δεν είναι αδιάφορο και όσοι έχουν αυτή την άποψη, ούτε και αυτοί μπορούν έτσι εύκολα να απορριφθούν. Η επέκταση των ιδίων πόρων ή ένας πανευρωπαϊκός φόρος δεν θα εξαφανίσει το πρόβλημα. Ένας λόγος για τον οποίο εγώ θα ήμουν κατά των διασώσεων, εάν ήταν η χώρη μου εντός της Ευρωζώνης, θα έλεγα πως οι διασώσεις αυτές δεν είναι πράξη γενεοδορίας. Αν ενδιαφέρονταν πραγματικά για τον Νότο η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα απελευθέρωνε τις χώρες αυτές από το ευρώ, την υπερτίμησή του και την λιτότητα, ανεργία και δυστυχία. Η ιδέα του κ. Κούν για τα διαφορετικά οράματα της Ευρώπης ήταν και πάλι ενδιαφέρουσα και εφάνταστη. Ακούγεται σαν ένα πατρονάρο τώρα, αλλά η ιδέα του νομίζω φορά εναλλακτικού και διαφορετικούς τρόπους προώθησης του ευρωπαϊκού εγχειρήματος και όχι απόρριψής του. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι μόνο έτσι, δεν έχω μια αυστηρά αγγλική ε, σκοπιά. Δεν απορρίπτω την Ευρώπη ως μια πολιτισμική οντότητα, αλλά απορρίπτω την Ευρωπαϊκή Ένωση με την ε, θέλησή της να δημιουργηθεί μια πολιτική οντότητα και όπου το μόνο ευρωπαϊκό θα είναι η γεωγραφία και δεν θα υπάρχει τίποτα το δημογραφικό ή πολιτισμικά, ε, δημογραφικά ή πολιτισμικά ευρωπαϊκό. Επιπλέον, με ενοχλεί το ότι η πολιτισμικα δημογραφικα η πολιτισμικα ευρωπαικο επιπλεον με ενοχλει το οτι η ευρωπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ταυτίζονται στα λόγια και όσοι είναι κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούνται κατά της Ευρώπης, ενώ δεν είναι. Η Ευρώπη σε αντίστοιχη με τι άλλε υπήρου, δεν είναι γεωγραφική ενότητα. Είναι ένα κομμάτι, το δυτικό κομμάτι της Ασίας γεωγραφικά. Οφείλεται λοιπόν η διαφορετικότητά της στους λαούς της και στους πολιτισμούς της. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάει για την ε, Ευρώπη και σκοπεύει να αντικαταστήσει με τον πολιτισμικό σχετικισμό και την δημογραφική αντικατάσταση. Σας ευχαριστώ, κύριος Γκουερέρο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να κάνω μερικά γενικά σχόλια για τις ομιλίες των καθηγητών Κουμ και Μαντζέλα. Και να αναφερθώ στα προβλήματα που αποτελούν την αιτία του μπλοκαρίσματος που παρατηρούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να επιληθούν πέραν των θεσμικών αλλαγών που θα γίνουν γιατί σχετίζονται με κάποιες συμπεριφορές που δείχνουν έλλειψη αλληλεγγύης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο καθηγητής Κουμ μίλησε εκτενώς για την αλλαγή της συμπεριφοράς ανάλογα με το αν πρόκειται για τη μεταφορά χρημάτων μέσω φορολογίας και ο μεταφοράς χρήματος μεταξύ μίας περιοχής και άλλης. Στην περίπτωση ε, χρημάτων από φορολογία ή μάλλον όταν έχουμε μεταφορές χρημάτων από εκείνους που, το έχουν, από εκείνους που έχουν προς εκείνους που δεν έχουν, είναι κάτι απολύτως νομιμοποιημένο ιδεολογικά, ακόμη και από μέλη της κεντροδεξιάς, όπως ο κ. Σασκόφσκι, ε, μεταξύ των, ε, η μεταφορά μεταξύ των εδαφών ε, είναι κάτι που μερικές φορές σχετίζεται και με την ητοπάθεια. Το βλέπουμε και στην ε, Ισπανία αυτό, στην πατρίδα μου. Αντί να επικρατήσει μια λογική ε, των ε, υψηλών εισοδημάτων που συμβάλλουν στην ευημερία των χαμηλών εισοδημάτων, έχουμε μια διαίρεση μεταξύ της περιφέρειας Α που καταλυστεύεται από την περιφέρεια Β ή από τις υπόλοιπες περιφέρειες. Αυτή η λογική φαίνεται ότι έχει επικρατήσει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την έναρξη της οικονομικής κρίσης. Υπάρχουν χώρες και οι κοινές τους γνώμες που θεωρούν ότι δεν θα πρέπει να είναι αλληλέγγυες με τα προβλήματα άλλων μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η κοινή γνώμη της μίας ή της άλλες χώρες έρχονται σε σύγκρουση και ουσιαστικά απαξιώνουν την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας τρόπος για να προχωρήσουμε είναι να αλλάξουμε την προσέγγισή μας ως προς το πρόβλημα. Η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις περιφέρειες είναι μια παρουσία οικονομικώς ισχυρή. Δεν μπορεί όμως να είναι ισχυρή η παρουσία αυτή όταν ο κοινοτικός προϋπολογισμός αντιστοιχεί μόνο στο 1% του ΑΕΠ, του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Επίσης, οι πόροι αυτοί, τα έσοδα αυτά, δεν προέρχονται από τις συνεισφορές των κρατών μελών που θεωρούν ότι είναι κυρίαρχοι του προπολογισμού, αλλά προέρχονται από τους φορολογούμενους, από τους πολίτες, μέσω του συστήματος των ιδιών πόρων, μέσω κάποιων φόρων και ούτω καθεξής. Βέβαια, εγώ δεν προτείνω κάποια ριζοσπαστική αλλαγή δηλαδή να περάσουμε σε, από την παρούσα κατάσταση σε μια τελείως διαφορετική κατάσταση ε, ιδιών πόρων ή να περάσουμε από το 1% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ στο 30% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Δεν προτείνω κάτι τόσο ρήξη και έλευθο, αλλά κατά τη γνώμη μου οι ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να αντιληφθούν την ε, πραγματική ωφέλεια της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και την θετική της επίδραση στην καθημερινότητά τους μέσω μιας ισχυρής οικονομικής παρουσίας στο κατάλληλο επίπεδο και να μην εκλαμβάνεται κάτι τέτοιο ως μεταφορά κονδύλιων από τη Γερμανία στην Ιταλία, από την Ολλανδία στην Ισπανία. Αλλά Ευρωπαίοι πολίτες να δείχνουν την ελεγγύη τους προς ένα κοινό σχέδιο και μέσω ενός κατάλληλου φορολογικού δημοσιονομικού συστήματος να πραγματοποιούνται μεταφορές ε, κονδυλίων, όπως γίνεται εντός ε, μιας χώρας, όπως γίνεται στο εσωτερικό του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως γίνεται στο εσωτερικό της Ισπανίας, προχωρώντας προς ένα σύστημα ιδίων πόρων. Δεύτερο σχόλιο αφορά τα τρία σημεία που μας ανέφερε ο κ. Μαντζέλα, την προσφυγή στο διεθνές δίκαιο προκειμένου να ε, ξεπεράσουμε το μπλοκάρισμα που υπάρχει στην Ένωση μεταξύ των χωρών. Αυτό όμω δεν μα εξυπηρετεί, γιατί έχουμε μια κοντόφθαλμη λύση, ψωμί για σήμερα και πείνα για αύριο, όπω λέμε στα Ισπανικά. Γιατί ουσιαστικά για να ξεφύγουμε από το προσωρινό μπλοκάρισμα, εκενώνουμε ε, τη γενετική μέθοδο από την ουσία τη προσφεύγουμε σε μια διακυβερνητική μέθοδο και, ένα, και το διεθνές δίκαιο που δεν είναι όμως το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο δεύτερο σημείο σας αναφερθήκατε στην εισβολή που γίνεται στο συνταγματικό δίκαιο των κρατών μελών. Και αυτή όμως είναι ε, μια αιτία της απώλειας νομιμοποίησης ε, που χάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις ε, διάφορες χώρες. Ο κύριος ο καθηγητής Μαντσέλα ε, γνωρίζει αυτή την κατάσταση, γιατί γνωρίζει τη συνταγματική εξέλιξη στην Ισπανία, ήταν αδύνατο να τροποποιηθούν για 35 ολόκληρα χρόνια κάποια στοιχεία του Ισπανικού Συντάγματο. Υπήρξαν πιέσεις για μερικές αλλαγέ. οι μερικές ήταν πιο σημαντικές από τις άλλες, αλλά είχαμε πολιτική απότελμα, δηλαδή πολιτικό μπλοκάρισμα, αδύνατο να γίνουν κάποιες αλλαγές. Εγκρίθηκε το Δημοσιονομικό Σύμφωνο και καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι χώρες θα πρέπει να εφαρμόσουν την δημοσιονομική ε, πειθαρχία στα συντάγματά τους και σε λιγότερο από μια εβδομάδα αναθεωρείται το Ισπανικό Σύνταγμα προκειμένου να, να περιλάβει και το σημείο αυτό. Οπότε εξέλιψε το επιχείρημα ότι μια συνταγματική αναθεώρηση προϋποθέτει ε, μια ορίμανση των προτάσεων, μια μεγάλη συνένεση, ευρεία συνένεση, ανάμειξη των πολιτών. Στην περίπτωση αυτή δεν συνέβη κάτι τέτοιο με το Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Οπότε αντιμετωπίζουμε αυτή την πίεση σήμερα. Μας λένε, αν αναθεωρήσετε το Σύνταγμα για να προσθέσετε την δημοσιονομική πειθαρχία μέσα σε μία εβδομάδα, για ποιο λόγο δεν μπορείτε να αναθεωρήσετε το Σύνταγμα και να προσθέσετε αλλαγές που εκκρεμούν στην Ισπανία εδώ και 30 χρόνια. Και τελευταία παρατήρηση, που δεν ξέρω είναι παρατήρηση παράπονα. Δεν έχουμε πολύ διαφορετικές εθνικές εμπειρίες. Δεν ξέρω σε τι σημείο φτάνουν αυτές οι διαφορές. Πάντως η σχέση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων δεν είναι σχέσεις ε, αδιάφθορης ε, αδελφότητας. Ε, κατά πάσα πιθανότητα και σε πολλές χώρες τα Εθνικά Κοινοβούλια φοβούνται ότι μία πρόοδο στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, οικοδόμηση θα αλλάξει το σχετισμό δυνάμεων και θα εκενώσει από αρμοδιότητες ή από ουσία τα εθνικά κοινοβούλια. Κάτι που ακούμε πολύ συχνά είναι ότι οι πολιτικές είναι όλο και πιο ευρωπαϊκές, ενώ η πολιτική είναι εθνικό ζήτημα. Είναι μια δυναμική που μας οδηγεί στο να λαμβάνουμε πολλές αποφάσεις εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση με συζητήσιμες, αμφισβητήσιμες από συνομιμότητα σε διαδικασίες, ενώ εκεί δηλαδή στις διάφορες χώρες γίνεται όλη η πολιτική συζήτηση περιώνουν σκιά ουσιαστικά γιατί δεν υπάρχει καμία συνέπεια, κανένα πρακτικό αντίκρισμα, αντίκρισμα αυτής της πολιτικής συζήτησης. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε και να ενισχύσουμε την δημοκρατική νομιμοποίηση αν δεν έχουμε ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα προέρχεται από εκλογές τις οποίες οι πολίτες θα γνωρίζουν τι αποφασίζουν και θα γνωρίζουν τη θέση όχι μόνο του Κοινοβουλίου αλλά και της κυβέρνησης. Και γι' αυτό και εγώ και η πολιτική μου ομάδα στο συνέδριο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών ε, αποφασίσαμε στην επόμενε εκλογέ να έχουμε ένα υποψήφιο που θα ταυτίζεται με την πολιτική μα οικογένεια. Και φαντάζομαι κάτι αντίστοιχο θα κάνουν και τα άλλα πολιτικά κόμματα. Νομίζω ότι έτσι θα πραγματοποιήσουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα. Οι πολίτες σε πολλές χώρες ψηφίζουν βουλευτές. Ξέρουν όμως ότι ανάλογα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα δημιουργηθεί η α ή β κυβέρνηση. Ενώ σήμερα, κατά τις ευρωεκλογέ, δεν υπάρχει αυτός ο συνειρμός και θα πρέπει να δημιουργηθεί αυτή η σχέση δηλαδή μεταξύ της ψηφοφορίας συγκεκριμένων ανθρώπων με τη διαμόρφωση μιας συγκεκριμένης πολιτικής κυβέρνησης. Αυτά και θα ήθελα να κλείδι να πω Κάτι που περιλαμβανόταν ε, μέσω στην παρουσίαση του καθηγητού Κουμ. Εγώ φυσικά είμαι υπέρ της Ευρώπης, είμαι ευρωπαϊστής, ε, πιστεύω ακράδαντα στην Ευρώπη και γνωρίζω ως Ισπανός ότι οι πρώτοι ε, που επηρέασαν το σύμφωνο σταθερότητας, οι πρώτοι που παραβίασαν το σύμφωνο σταθερότητας δεν ήταν οι χώρες του Νότου, και μάλιστα τότε οι χώρες του Νότου έδειξαν μεγάλη ελληνική προς τη Γερμανία που ήταν εκεί η χώρα που παραβίασε το Σύμφωνο Σταθερότητας. Και μάλιστα κάποια προβλήματα του τραπεζικού κλάδου που παρατηρήσαμε στη χώρα του Νότου οφειλόταν σε ε, ελλείμματα στο εμπορικό ισοζύγιο και στο ισοζύγιο πληρωμών εξαιτία της ροής κεφαλαίων από το Νότο προς το Βορρά και αυτή τη στιγμή ο Βορράς χρηματοδοτείται δωρεάν ενώ ο Νότος χρειάζεται να πληρώσει για τη χρηματοδότηση ε, υπέρογκα επιτόκια 6% μερικές φορές και αυτή την κατάσταση δεν θα την είχαμε σε, μια, σε ένα ομόσπονδο φεντεραλιστικό κράτος. Και καλό θα ήταν να την αποφεύγαμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όποιος και είναι ο βαθμός του φεντεραλισμού που θα εφαρμόζει αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στους καθηγητές για να απαντήσουν. Και πρώτα εκείνοι που μίλησαν το πρωί, πάντα στη δεύτερη ενότητα και μετά εκείνοι που μίλησαν το απόγευμα, στην τρίτη. Δυστυχώς ε, έχουμε περιορισμένο χρόνο, ένα πεντάλεπτο για τη δευτερολογία σας ε, παρακαλώ να τον τηρείτε με τη σειρά που θέλετε εσείς. Θα μπορούσαμε όμως να δώσουμε με τη σειρά το λόγο ε, με τη σειρά που μιλήσατε το πρωί. Ο καθηγητής ο κύριος Δεούς, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δύο σχόλια θα κάνω μόνο. Αυτά που άκουσα στη συζήτηση. Το πρώτον είναι αυτή η ιδέα πως η πολιτικοποίηση είναι αναγκαία και επιθυμητή και το αντιλαμβάνομαι αλλά εγώ θα ήθελα να τονίσω πως κατά κάποιο τρόπο ήδη συμβαίνει όχι όπως το περιμέναμε όμως συμβαίνει. Γιατί αν δείτε τις εκλογές που έλαβαν χώρα σε ευρωπαϊκές χώρες φέτος, σαφώς ήταν ευρωπαϊκές. Τι εννοώ δηλαδή. Οι εκλογές στην Ελλάδα ε, περιστρέφονταν γύρω από το τι σημαίνει το να είναι κανείς μέλος ε, στο ευρώ και τη σχετική πειθαρχία. Οπότε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι και ε, στις Ολλανδικές εκλογές ε, ήταν ζήτημα το να είναι η χώρα ή όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έπαιξαν ρόλο και στις γαλλικές προεδρικές εκλογές τα, τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Αυτό δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Γιατί, γιατί ε, ο τρόπος με τον οποίο συνέβη Ας πάρουμε παραδείγματος χάρη το γαλλικό παράδειγμα το οποίο γνωρίζω καλύτερα. Ο τρόπος αυτός δεν ε, συμβαζόταν με αυτό το οποίο σκεφτόμαστε όταν λέμε κάποιες εκλογές ε, ευρωπαϊκές. Δηλαδή δεν υπήρχε η σύγκρουση μεταξύ φεντεραλιστών και μη. Ε, ήταν τα ζητήματα αυτά τα οποία ανέφερε και ο κύριος Τρασκόφσκι, δηλαδή δουλειές, απασχόληση, οικονομία, μετανάστευση. Όχι το εάν θέμα Ομοσπονδιακή Ένωση ή όχι. Αλλά γνωρίζοντας πως οποιαδήποτε πολιτική θέλει κανείς να ακολουθήσει σε σχέση με αυτά τα ζητήματα, ε, κρίνεται σε μεγάλο βαθμό από το τι κάνει και θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε, όσοι κατεβαίνουν στι εκλογέ. δεν πρέπει να πούν μόνο το τι θα κάνουν εάν ε, βγουν αρχηγοί κράτου ε, ή κυβερνήσεων αλλά και το τι θα κάνουν στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Κάποιοι θα έλεγαν πως αυτό είναι καλό γιατί πολιτικοποιεί τη συζήτηση για την Ευρώπη και ως ένα βαθμό είναι σωστό. Έχω όμως κάποιους φόβους. Τι εννοώ. Αν δεν υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα κομμάτων, είναι, αυτό το οποίο έχουμε είναι μια πόλωση, όπου ο κόσμος από τον Νότο θα εκφράζει τα προβλήματα που έχει με τους βόρειους ας πούμε συμπατριώτες τους στην Ένωση και οι άνθρωποι από το βορρά θα εκφράσουν τη δυσπιστία τους για τους νότιους κτλ. κτλ. Και το λέω αυτό για δύο λόγους. Πρώτον για να πω πως η πολιτικοποίηση έχει ξεκινήσει και το πραγματικό ερώτημα είναι εάν θέλουμε να μην απειληθεί η σταθερότητα της Ένωσης μπορούμε να έχουμε αυτό να αποτελέσει ένα σοβαρό κίνητρο για περαιτέρω πολιτικοποίηση των ευρωεκλογών. Αλλά, εδώ είναι το πρόβλημα και η δεύτερη παρατήρησή μου, η πολιτικοποίηση των ευρωεκλογών σημαίνει ακριβώς να εστιάσουμε στα ζητήματα που έχουν σημασία για τους πολίτες. Δουλειές, απασχόληση, οικονομία, μετανάστευση. Δείτε μας αρέσει ή όχι. Και αυτό προϋποθέτει όχι μόνο το ότι τα κόμματα θα θελήσουν να παίξουν το παιχνίδι αλλά και την δυνατότητα να έχουν αποτελέσματα γιατί τα ζητήματα αυτά που αφορούν τους πολίτες είναι ζητήματα αποτελεσμάτων αλλά αποτελέσματα για τα οποία η Ένωση ίσως να μην έχει όλα τα μέσα τα οποία θα χρειαζόταν για να αντιδράσει. Όπως είπαμε, ο προπολογισμός είναι στο 1% του ΑΕΠ και δύσκολα μπορεί κανείς να αντιληφθεί πώς μπορεί να έχει ε, μια λογική μακροοικονομική πολιτική, έτσι για να φέρω ένα παράδειγμα. Οπότε είναι δύσκολο να δούμε πώς οι ρυθμιστικές αρμοδιότητες της Ένωσης ε, θα αρκέσουν για να ανταποκριθούν στις ανησυχίες των πολιτών. Οπότε, αν ακολουθήσουμε τη λογική αυτή μέχρι τέλους, πρέπει να ρωτηθούμε μήπως η πολιτικοποίηση των ευρωπαϊκών εκλογών μας οδηγήσει στο να ξαναδούμε την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Ένωσης και κρατών μελών. Και το λέω αυτό γιατί θεωρώ πως δεν θα είμαι ο μόνος που ε, βλέπει μια τέτοια λογική. Και βεβαίως στο μυαλό πολλών θα αποτελέσει ένα καλό λόγο για να μην πάμε στην κατεύθυνση πολιτικοποίηση. Βεβαίω πολλοί λένε πώ έρχεται, θα γίνει, τα μεγάλα κόμματα έχουν αποφασίσει να γίνει αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εγώ θα περιμένω. Υπάρχει μια ωραία βρετανική παροιμία που λέει πως οι γαλοπούλες δεν ψηφίζουν τα Χριστούγεννα, υπέρ των Χριστουγέννων δηλαδή, Οπότε δεν ξέρω εάν εθνικά κόμματα θα παίξουν θετικό ρόλο στην πολιτικοποίηση αυτή. Ας ε, ελπίσουμε όμως πως θα αποτυχθώ λάθος. Ευχαριστώ. Μου φαίνεται ότι ο καθηγητής Βέσελς α, δεν θέλει να μιλήσει. Ωραία, θα δώσουμε το λόγο τότε στον καθηγητή κύριο Βάιλα. Uh, να σας ευχαριστήσω για τα σχόλιά σας. Και δεν νομίζω πως τα ζητήματα τα οποία έτεθησαν μπορούν να απαντηθούν έτσι με σλόγγαν. Λίγα λόγια για τον Δήμο βεβαίω. Ε, ε, εγώ πάντα έλεγα πως όταν μιλάμε για Ευρωπαϊκό Δήμο δεν πρέπει να σκεφτόμαστε Ευρωπαίους όπως λέμε Γάλλοι, Άγγλοι, Ιταλοί. Είναι ένα Δήμος που θα οικοδομηθεί γύρω από τις αξίες και την αλληλεγγύη αντί για οποιαδήποτε έτσι πιο φυσική σχέση. αυτό και βεβαίως ε, μια οικαιότητα η οποία θα οικοδομηθεί μεταξύ των διαφόρων μερών της Ευρώπης και νομίζω πως μπορεί να παραμείνει η μοναδικότητα του ευρωπαϊκού οικοδομήματος που διατηρεί κυρίαρχα κράτη-μέλη αλλά έχει και μεγάλο βαθμό ολοκλήρωσης από την άλλη και να ε, σκεφτούμε αυτά τα οποία είπε ο κύριος ε, Κούν και ο κύριος Ντεούς η πολιτικοποίηση είναι σημαντική Δηλαδή να έχουμε επίσημες δομές αλλά να μην έχουμε πολιτική, να μην έχουμε αντιπαράθεση. Οπότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μια κρίση ταυτότητας. Είναι το θεσμικό όργανο που αναζητά συμβασμού στα περισσότερα ψηφίσματα είναι διακομματικά με κέντρο αριστερά και κέντρο δεξιά αυτό είναι καλό για την Ευρώπη υπό την έννοια πως προωθεί διάφορα θέματα αλλά χάνουμε έτσι το ενδιαφέρον του λαού Οπότε πρέπει να γίνει εδώ μια επαρξιακή επιλογή. Η πολιτική δεν είναι διαφωνία για τη διαφωνία, αλλά διαφωνία και επιλογή. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο πρέπει να γίνει το μέρος εκείνο όπου ο κόσμος όπου δεν είναι ικανοποιημένος με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ακούει τη φωνή του και θα εκπροσωπείται με τρόπο ουσιαστικό και μπορούν να υπάρξουν μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ κέντρο αριστεράς και κέντρο δεξιάς. Οπότε πρέπει εδώ πέρα δηλαδή να δούμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη και για πολλές δεκαετίες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρούσε αυτόν ε, το υπεύθυνο θεσμικό όργανο που αναζητούσε το συμβιβασμό και ήταν επιτυχημένο αλλά βεβαίως έχασε την ελκυστικότητά του. Είναι δύσκολο για οποιοδήποτε ευρωβουλευτή να πει να βάλει το χέρι στην καρδιά και να πει πως ε, επανεξελέγει ε, με βάση τα όσα έκανα και πέτυχα στο κοινοβούλιο και είπα στο κοινοβούλιο. Γιατί ακριβώς δεν υπάρχει η αρχή αυτή της επανεκλογής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτή είναι η ουσία της πολιτικής και η ουσία της δημοκρατίας. Οπότε θεωρώ πως δεν χρειάζεται έτσι γρήγορες λύσεις, αλλά ένας ε, αναπροσανατολισμός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει με τρόπο ουσιαστικό και όχι συνθήματα να ξανααποκτήσει αυτή την έννοια του Vox Populi. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καθηγητά. Και τώρα ο καθηγητής κ. Σκούμ. Μια πολύ σύντομη παρατήρηση μόνο. Θα αναφερθώ σε ένα και μόνο ζήτημα. Και αυτό είναι ο ισχυρισμό ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να συνδέεται με το λαό ή τους λαούς με τον τρόπο που συνδέονται εθνικά κοινοβούλια και εθνικά κόμματα, διότι τα θέματα εδώ που διαπραγματεύεται το κοινοβούλιο δεν είναι θέματα που αγγίζουν τον κόσμο, ο κόσμος ότι ε, τον αφορούν. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Είναι πραγματικά μεγάλη έκπληξη. Ο Στάινμπροκ που τώρα διορίστηκε υποψήφιο των σοσιαλδημοκρατών για την καγκελαρία, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να κατεβάζει ένα έγγραφο για τον τραπεζικό τομέα και τη μεταρρύθμιση. Και τι λέει το έγγραφο αυτό, τι προτείνει. Αυτά που ήδη συζητούνται εδώ και καιρό και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και εδώ στο Κοινοβούλιο. Παράδειγμα, ε, την οδηγία για την εξυγίανση των τραπεζών ή μια ιδέα που είναι απλώς στη συζήτηση και δεν έχει γίνει πρόταση, ε, το να γίνει ένας διαχωρισμός της ε, τράπεζες, ε, τις δραστηριότητε υψηλού κινδύνου από τις καταθέσεις κτλ. Ε, όλα αυτά ε, είναι αντικείμενο συζήτησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά κανείς δεν ακούει τις συζητήσεις αυτές, ούτε παρακολουθεί πώς διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο, στα εθνικά μίντια. Μόνο όταν το κάνει ζήτημα ένας πολιτικός στη χώρα του. Αλλά όταν τα συζητάει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ενδιαφέρεται κανεί. Και αυτό είναι πρόβλημα και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα πρέπει να σκεφτείτε πώ θα το αντιμετωπίσετε, πώ θα το ε, διορθώσετε αυτό ε, για να παίξει το ρόλο που του αξίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ και τώρα ο καθηγητής Ματζέλα, αν θέλει και θεωρεί σκόπιμο να απαντήσει. Είναι γεγονός ότι πλέον δεν υπάρχει καμιά διαφορά, δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά και εθνικά ζητήματα, δεν είναι διακριτά αυτά. Ακριβώς αυτό το λόγο θα ήταν αυτοκτονικό στις επόμενες ευρωεκλογές ε, ε, να κατατεθούν ίδιοι μηχανισμοί με τις εθνικές αντιπροσωπείες προς ψήφιση στον Ευρωπαίο πολίτη, ό,τι έχουμε μέχρι τώρα, δηλαδή και ο τρόπος με τον οποίο εκλέγεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από το 2014 ε, θα πρέπει να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Όπως είπα και προηγουμένως, να απεθνικοποιηθούν οι ευρωεκλογές, να γίνουν ευρωπαϊκές. Δεν λειτουργεί πια αυτό το σύστημα. Και πλέον αυτό ε, δεν είναι μόνο υποχρέωση, ε, ε, μάλλον υποχρέωση και περισσότερο από ό,τι ανάγκη. Υπάρχει πολιτικοποίηση λέτε. Δεν είναι μόνο αυτό. Θα πρέπει να βρούμε ένα μηχανισμό που να δίνει μια φωνή, ναι, μια πολύ ισχυρή φωνή που ακούγεται σήμερα είναι οι αντιευρωπαϊστές και ευρωσκεπτικιστές. Θα πρέπει και εμείς κάπως να το αντιμετωπίσουμε αυτό από την άλλη πλευρά. Για να υπάρχει λοιπόν αυτή η απεθνικοποίηση και να ε, ψηφιστούν πραγματικά Ευρωπαίοι βουλευτές και όχι με κριτήρια εθνικής πολιτικής, να έχουν μια πραγματική ευρωπαϊκή εντολή δηλαδή ε, και να έχει και ένα αποτέλεσμα αυτό που μας ενδιαφέρει και αυτό θα πρέπει να προταθεί στους ε, εκλογείς το 2014 ε, γίνεται μεγάλος λόγος για την πολιτική ένωση πολύ κακό για το τίποτα Τι, ποια είναι η πολιτική ένωση αυτή δεν είναι κάτι που συνδέεται με τους μηχανισμούς με το εκλογικό σώμα πώς γίνεται αυτό τι είναι αυτά χτίσματα στην άμμο είπε ο βουλευτής Γκερέρο ότι επί μία τριαντακονταετία το Ισπανικό Σύνταγμα ε, δεν άλλαξε καθόλου και σε 15 μέρες ε, αμέσως ως διαμαγές. Το άρθρο 4, παράγραφος 2, αναφέρεται στο σεβασμό της συνταγματικής ταυτότητας των κρατών και πλέον αυτό το αντιλαμβανόμαστε ε, με μια ε, πιο ευρία έννοια. Ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διευρυνθεί η έννοια της συνταγματικής οντότητας για να μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα και αυτές οι αντιφάσεις. Σε ό,τι αφορά την διακοινοβουλευτική συνεργασία, όπως και στο γάμο, εντάξει, προξενιό είναι, αλλά δύο πρέπει να συνενέσουν για να γίνει αυτός ο γάμος. Μέχρι τώρα εγώ δεν έχω αισθανθεί από τις πρωτοβουλίες αυτές και για το Δημοσιονομικό Σύμφωνο ας πούμε θα δείξει ε, η εξέλιξη αλλά δεν έχω δει ακόμα πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που λέει στο άρθρο 13 Δημοσιονομικό Σύμφωνο, διάσκεψη. Ε, έρχονται λοιπόν οι αρμόδιες επιτροπές από τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και καλή την πίστη ζητούμε. Αυτά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μαντζέλα, καθηγητά. και ε, ε, ήσασταν και ευρωβουλευτής, δεν χάνετε αυτό τον τίτλο. Ε, και περνούμε στην επόμενη ενότητα, η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση πέραν των υφισταμένων μηχανισμών. Ίσως είναι και το πιο ενδιαφέρον αυτό. Και θα παρακαλέσω τον καθηγητή Τζαν Λουίζη Τοσάτο να έρθει εδώ στο Προεδρείο ο καθηγητής στο ΖΑΤΟ διδάσκει διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο στο Πανεπιστήμιο Λασεπιέντσα της Ρώμης. Είναι μέλος διαφόρων ε, διεθνών θεσμών και ε, συγγραφέας πολλών ε, συγγραμμάτων για το διεθνές, δημόσιο και ιδιωτικό δίκαιο. Παρακαλώ καθηγητά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά πως οι απογευματινές συνεδριάσεις και τα σεμινάρια είναι δύσκολα, ειδικά αν είναι και το δεύτερο μέρος ε, της απογευματινής συνεδρίασης. Οπότε θα προσπαθήσω να είμαι όσο ε, το δυνατόν πιο σύντομος. Το θέμα μας λοιπόν είναι πέραν από τους υφιστάμενους μηχανισμούς και όπως αναφέρατε κύριε Πρόεδρε Α, μάλιστα, κατάλαβα. Ευχαριστώ. Όπως αναφέρατε, λοιπόν η συζήτηση κάλυψε πολλές από τις πτυχές ε, του θέματος. Ήδη λοιπόν έχει συζητηθεί το τι μπορεί να γίνει για να πάμε πέρα από τους υφιστάμενους μηχανισμούς. Εγώ θα ήθελα να επικεντρωθώ στο θέμα το οποίο βλέπετε εκεί απέναντι στη διαφάνεια Δηλαδή πώς θα βελτιωθεί ο μηχανισμός ευελιξίας ε, εντό του ευρωπαϊκού δικαίου. Πάρα πολλά συζητήθηκαν σήμερα το πρωί για την ευελιξία εντός του ευρωπαϊκού δικαίου και εκτός του ευρωπαϊκού δικαίου. Και θεωρώ πως σωστά υπόθηκε πως ε, η ευελιξία εντός του ευρωπαϊκού δικαίου, οι διεθνείς συμφωνίες εκτός του ευρωπαϊκού δικαίου είναι κάτι το θεμητό, αυτό συζητήθηκε και πιθανότατα αναγκαίο όταν δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα για να προωθηθεί η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση αλλά ταυτόχρονα θα ήταν πολύ πιο χρήσιμο ε, για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ακόμα και υπό μορφή μιας διαφορετικής ολοκλήρωσης να ε, συμβεί κάτι τέτοιο εντός του πλαισίου του ευρωπαϊκού δικαίου και όχι εκτός. Οπότε τι μπορεί να γίνει για να βελτιώσουμε τα μέσα της ευελιξίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικαίου έτσι ώστε στο μέτρο του δυνατού οποιασδήποτε νέες εξελίξεις να ενταχθούν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικαίου. Αυτό λοιπόν θα προσπαθήσω να αναπτύξω. Τρεις λοιπόν προτάσεις έχω να κάνω. Πρώτον, να εισαχθεί ευελιξία στο επίπεδο του πρωτογενούς δικαίου, των συνθήκων, δεύτερον να αυξήσει ευελιξία στο επίπεδο του δευτερογενούς δικαίου και τρίτον να υπάρξει μία ρήτρα εξόδου για όλες τις ευέλικτες πρωτοβουλίες. Να ξεκινήσω με το πρώτο λοιπόν. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ευελιξία στο επίπεδο του πρωτογενούς δικαίου. Ξέρετε πως η αναθεώρηση των συνθήκων είναι αυτή που είναι τώρα με τη συνθήκη της Λισαβόνας υπάρχει μια απλοποιημένη διαδικασία αναθεώρησης ούτως ή άλλως είτε μιλάμε για την ε, τακτική διαδικασία είτε για την απλοποιημένη διαδικασία χρειάζεται ομόφωνη κύρωση από όλα τα κράτη-μέλη οπότε αυτό σημαίνει μια ακαμψία για οποιαδήποτε τροποποίηση του πρωτογενούς δικαίου εντός ένωμης τάξης της Ένωσης. Είναι λοιπόν φυσιολογικό για οποιοδήποτε σύνταγμα να προβλέπει μια πιο δίσκαμπτη διαδικασία αλλαγής. Αλλά εδώ έχουμε απόλυτη ακαμψία γιατί είτε υπάρχει ομοφωνία μεταξύ όλων των κρατών μελών είτε δεν υπάρχει αναθεώρηση. Οπωσδήποτε Ισχύει αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι κράτος. Βασίζεται σε συνθήκες. Οι συνθήκες δεν είναι σύνταγμα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πολύ άκαμπτο το σύστημα. Ποια θα μπορούσε να είναι η αλλαγή λοιπόν που θα μπορούσαμε να προτείνουμε. Κατά την άποψή μου δεν είναι εφικτό να σκεφτούμε μία διαδικασία με την οποία με μια ισχυρή πλειοψηφία μπορεί να γίνει αλλαγή των συνθήκων με δεσμευτικό αποτέλεσμα και για τις χώρες οι οποίες δεν ε, συνενούν. Δεν νομίζω πως έχουμε φτάσει εκεί ε, σε, τουλάχιστον στον παρόν στάδιο ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης αλλά αυτό το οποίο θα μπορούσε να γίνει είναι να πούμε σύμφωνα με το μηχανισμό ευελιξίας να πούμε πως ε, η αλλαγή των συνθήκων μπορεί να γίνει με δεσμευτικό αποτέλεσμα για τις χώρες που την έχουν κυρώσει. Και ίσως θα ήταν υπερβολικό να εισαχθεί μια τέτοια αλλαγή για οποιαδήποτε αλλαγή τη συνθήκη, αλλά θα μπορούσαμε να σκεφτούμε παραδείγματο χάρη την απλοποιημένη διαδικασία αλλαγής των συνθήκων που περιορίζεται σε συγκεκριμένες ε, πολιτικές. Θα ήταν εφικτό να πούμε πως σε σχέση με αυτές τις αλλαγές μπορούν να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις για τις χώρες οι οποίες κυρώνουν, ακόμα και αν δεν υπάρχει ομοφωνία, αλλά θα ισχύσει για τις χώρες οι οποίες έχουν, την έχουν κυρώσει και υπό την προϋπόθεση μιας συγκεκριμένης ε, πλειοψηφίας των κρατών Να σας δώσω ένα παράδειγμα. η αλλαγή που έγινε στο άρθρο 136 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχει ακόμα τεθεί εν ισχύ αλλά θα ισχύσει σύντομα. Η τροποποίηση αυτή επηρεάζει μόνο τις χώρες που ανήκουν στην Ευρωζώνη αλλά η θέση ενισχύει των αλλαγών της συνθήκης είναι υπό την αίρεση της κύρωσης από όλα τα κράτη μελικά, το οποίο βεβαίως είναι παράδοξο. Γιατί δεν είναι προφανές το γιατί μια τροποποίηση η οποία απευθύνεται μόνο σε κάποια κράτη-μέλη, στην περίπτωσή μας τα κράτη-μέλη που είναι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι υπό την αίρεση της έγκρισης των κρατών μελών που δεν ε, θα τους αφορά αυτή η αλλαγή. Οπότε, θα πρότεινα εγώ να εισαχθεί αυτή η αλλαγή συνθήκη. Γνωρίζω πως είναι αλλαγή της συνθήκης. Και άρα πρέπει να περάσει αναθεώρηση της συνθήκης, αλλά είναι μία μικρή αναθεώρηση που θα δώσει στην ένωμη τάξη της Ένωσης την δυνατότητα να εισαχθεί μια ευελιξία στο επίπεδο του πρωτογενούς δικαίου που αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται. Η δεύτερη μου πρόταση, εκεί είμαι ακόμα, αυτό το περάσαμε Yeah, no, that's, uh, that's too much. Okay, so my second proposition is... Uh, η δεύτερη μου πρόταση είναι να αυξηθεί η ευελιξία στο επίπεδο του δευτερογενούς ε, δικαίου, όπου υπάρχει ήδη κάποια ευελιξία. Έχουμε γνωστά μέσα την ενισχυμένη συνεργασία και το άρθρο 136. Υπάρχει και κάτι άλλο. Η δομημένη συνεργασία στο πλαίσιο της άμυνας, αλλά ε, τα δύο βασικά γενικά μέσα που επιτρέπουν την ευελιξία στο επίπεδο του δευτερογενούς δικαίου είναι αυτά τα οποία ανέφερα πριν, δηλαδή άρθρο 136 για τις χώρες της Ευρωζώνης και ενισχυμένη συνεργασία για τις χώρες εκείνες που ε, συμμετέχουν σε μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Θεωρώ λοιπόν πως η σχετικά περιορισμένη χρήση που έχει γίνει ε, αυτή τη στιγμή των δύο αυτών μέσων οφείλεται στο ότι Ε, τα μέσα αυτά είναι κάπως δυσκίνητα και βαριά. Ας δούμε παραδείγματος χάρη την ενισχυμένη συνεργασία η οποία απαιτεί έναν αριθμό διαδικαστικών προϋποθέσεων έναν αριθμό ουσιαστικών προϋποθέσεων και θεωρώ πως κάποιοι από αυτούς μπορεί να απλοποιηθούν και συγκεκριμένα αυτό αφορά την ομοφωνία που απαιτείται για να δοθεί η άδεια για ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και στο πως υπάρχει μονοπόλιο της Κομισιόν για οποιαδήποτε πρωτοβουλία. Γιατί οποιαδήποτε πρωτοβουλία ενισχυμένης συνεργασίας δεν μπορεί να ξεκινήσει χωρίς ε, πρόταση της Κομισιόν. Εάν αυτά τα δύο στοιχεία, αυτοί οι δύο όροι χαλαρώσουν, θεωρώ πως η ενισχυμένη ε, συνεργασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί περισσότερο από ότι στο παρελθόν. Σημειώνω πως στο δημοσιονομικό σύμφωνο τα κράτη τα οποία συμμετέχουν έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να χρησιμοποιήσουν περισσότερο την ενισχυμένη συνεργασία. Επίσης, έχουν αναφέρει πως θέλουν να χρησιμοποιήσουν περισσότερο το άρθρο 136. Οπότε, αυτό το οποίο θα έλεγα είναι το πώς θα βελτιωθεί η χρήση του άρθρου 136. Εδώ πέρα λοιπόν θεωρώ πως το άρθρο 136 έχει αυτή τη στιγμή περιορισμένο πεδίο εφαρμογής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάποιους ε, σκοπούς, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να λύσει όλα τα προβλήματα τα οποία ε, σχετίζονται με τη δημιουργία αυτού του οποίου λέμε μιας ε, πραγματικής οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Ε, συζητήθηκε σήμερα το πρωί πως ε, δεν είναι ε, το άρθρο 136 δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά περισσότερων αρμοδιοτήτων για να χρησιμοποιηθεί μια πραγματική δημοσιονομική και οικονομική ένωση δηλαδή για να δημιουργηθεί ένας νέος προϋπολογισμός μια νέα δημοσιονομική αρμοδιότητα η αρμοδιότητα δαπανών ή φορολογίας. Για να γίνει αυτό πρέπει να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 136. Αλλά αυτό ε, θα πρέπει, μπορεί να είναι σχετικά απλό. Όπως σχετικά απλή ήταν η τροποποίηση του άρθρου 136 που ήδη ξεκινήσει. επί τη Είναι κάπως παράδοξο το ότι μετά την τροποποίηση του άρθρου 136 και της νέας παραγράφου 3 καταφύγαμε σε μια συνθήκη εκτός του ευρωπαϊκού δικαίου γιατί μόλις ε, έγινε ε, η τροποποίηση θα ήταν λογικό να γίνει κάτι εντός του ευρωπαϊκού δικαίου και της ευρωπαϊκής ενόμης τάξης και όχι εκτός και το πεδίο εφαρμογής της νέας αυτής αλλαγής θα ήταν πάλι οποιαδήποτε νέα εξέλιξη να ενταχθεί εντός της, ε, ένομης, της ευρωπαϊκής τάξης. είμαι σύντομο τώρα για το τρίτο μου σημείο. Thank you. It's... Ε, and it is the question of... Ναι το ζήτημα λοιπόν της εξόδου. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ ακριβείς οι πρόνοιες της ε, συνθήκης όσον αφορά βεβαίως ε, την ε, ένταξη σε μία, στην πρωτοβουλία της ευελιξίας. Γιατί και λογικό είναι να λέμε πως δεν υπάρχει διάκριση όσον αφορά την ένταξη σε μία νέα α, πρωτοβουλία. Λογικό αυτό. Αλλά από την άλλη, η συνθήκη δεν λέει τίποτα για το ζήτημα της εξόδου. Τώρα υπάρχει μία ρήτρα για την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν υπάρχει διάταξη για την έξοδο από κάποιο υποσύνολο της Ευρωπαϊκής Ενόμης Τάξης. Και θεωρώ πως δεν θα ήταν άστοχο να εισαχθεί ένα ειδικό καθεστώς το οποίο θα ρύθμιζε αυτό το θέμα. Είναι γνωστό πως αυτό συζητιέται σε σχέση με την ε, νομισματική ένωση, το ευρώ. Είναι δυνατόν να βγει κανείς από το ευρώ. Είναι δυνατόν να βγει μόνο από το ευρώ ή πρέπει να βγει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ πως θα ήταν λογικό να εισαχθεί εδώ πέρα κάτι το πιο συγκεκριμένο και θεωρώ πως πρέπει να σημειώσουμε πως στην ε, πρόσφατη απόφαση του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου υπάρχει μια παράγραφος στην οποία το δικαστήριο ασχολείται με το πρόβλημα της εξόδου από τη συνθήκη του μηχανισμού σταθερότητας όπου λέει πάλι πως δεν υπάρχει κάποια διάταξη που θα δώσει τη δυνατότητα σε μια χώρα να βγει από τη συνθήκη. Αλλά αυτό είναι δυνατόν ε, με βάση το γενικό διεθνέ δίκαιο γιατί ε, είναι αναγκαίο βεβαίω να υπάρχει δυνατότητα εξόδου. Αλλά οπωσδήποτε οι γενικοί κανόνε του διεθνούς δικαίου ε, μπορούν να ισχύσουν αλλά περιορίζονται σε κάποιους περιπτώσεις και πιο συγκεκριμένοι κανόνες ε, που θα δημιουργούσαν ένα καθεστώς εξόδου θα ήταν καλή για τις πρωτοβουλίες αυτές της ευελιξίας της λεγόμενες γιατί θα διευκόλυναν και την είσοδο σε, σε ένα καθεστώς ευελιξίας δηλαδή να υπάρχει και δυνατότητα εξόδου Ευχαριστώ Ευχαριστώ και θα περάσουμε τώρα στην καθηγήτρια Βιβιάν Σμιτ που διδάσκει στην έδρα Ζαμονέ για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, καθηγήτρια διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Βοστόνης, πρώην διευθύντρια της Ένωσης για τις Ευρωπαϊκές Σπουδές στις Ηνωμένε Πολιτείε. Έχει ήδη λάβει θέση η κυρία Σμιτ και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Μου ζητήσατε να μιλήσω για την διαφοροποιημένη ολοκλήρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ρόλο της ε, ευρωπαϊκής πολιτικής οικονομίας. Εγώ θα αναφερθώ και στη σημερινή συζήτηση, την πρωινή. Ε, θα μιλήσω για κάποια γενικά θέματα, ζητήματα δημοκρατίας, ε, θεσμών, αλλά και την πολιτική οικονομία. Θα ξεκινήσω με την πραγματικότητα της διαφοροποιημένης ολοκλήρωσης. Συνεχίζοντας αυτά που μας παρουσίασε το πρωί Γιάννης Αμανουηλίδης, θα μιλήσω για το πρόβλημα της δημοκρατίας, μετά από αυτά που ακούσαμε από πολλούς και ιδιαίτερα από τον καθηγητή Βάιλερ, θα μιλήσω για το πρόβλημα που έχει η ευρωπαϊκή πολιτική χωρί, οι ευρωπαϊκές πολιτικές χωρίς πολιτική και η, ευρωπαϊκή, η εθνική πολιτική χωρίς πολιτικές. Και το θέμα είναι πώς ε, μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να συγκεντρώσει και την πολιτική και τις πολιτικές. Επίσης θα υποβάλω κάποιες προτάσεις για το τι μπορούμε να κάνουμε για την ευρωπαϊκή πολιτική οικονομία που εξαρτάται φυσικά και σε περισσότερη νομιμοποίηση και δημοκρατία. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα να αναγνωρίσουμε την πραγματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εμπεριέχει μεγάλο βαθμό διαφοροποιημένης ολοκλήρωσης ήδη. Ποτέ δεν πρόκειται να γίνει ένα ομόσπονδο υπερκράτος, οπότε ε, ας σταματήσουμε να ανησυχούμε για το θέμα αυτό. Ούτως ή άλλως ε, θα έχουμε ε, δύο ταχυτήτων Ευρώπη και τώρα και στο μέλλον. Αλλά δεν θα πρέπει να έχουμε μια αντιπαράθεση σκληρού πυρήνα και περιφέρειας, ούτε επιλεκτική Ευρώπη, Ευρώπη à la carte. Ε, θα είναι περισσότερο μια περιφερειακή ένωση ε, χωρών εθνών που έχουν συμπεριληφθεί σε μια ευρύτερη ένωση. Θα μπορούσαμε πούμε και ομοσπονδία ε, κρατών εθνών, αν όχι όπως την είπα εγώ, όπως είπε ο Παρόσο. Και αντί να έχουμε ένα σκληρό πυρήνα, θα μπορούσαμε να έχουμε έναν χαλαρό πυρήνα μεγάλου αριθμού χωρών που συμφωνούν για κάποιες ε, πολιτικές ε, αλληλοεπικαλυπτόμενες. Αυτό που μας ε, παρουσίασε το πρωί ο Γιάννη. Και αυτό είναι σημαντικό για να αντιληφθούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ω οντότητα που επιτρέπει τη διαφοροποίηση, αλλά εξασφαλίζει και περισσότερη ολοκλήρωση με ένα ενιαίο πλέγμα θεσμών, με πολλέ κοινοτικέ πολιτικέ και όπως είπαν κάποιοι προλαλήσαντες και με μεγάλο βαθμό και ενισχυμένη συνεργασία. Χρειάζεται όμως κάποιες μεταρρυθμίσεις για να συμβούν όλα αυτά. Και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά του ε, θεσμικού κανόνε. Υπάρχει πρόβλημα με τον κανόνα τη ομοφωνία. Προτιμούμε ενισχυμένε πλειοψηφίε, 4 πέμπτων, με ρήτρε αυτοεξαίρεση. Είναι ε, κάπως, ήταν κάπως ειρωνικό αυτό που είπε ε, ότι ε, αμέσως ο, ο Κάμερον το νομοποίησε με το βέτο του για το δημοσιονομικό σύμφωνο πρόκειται για την απαρχή ουσιαστικά ε, ε, υπερπλειοψηφιών, πραγματικές υπερπλειοψηφίες, δηλαδή με μόνο με μία, μόνο με μία αυτο, αυτοεξαίρεση. Και αν συμφωνούσαν σε αυτό τα κράτη-μέλη, δεν θα χρειαζόμασταν καν να θεώρηση της συνθήκης. Οπότε διαφυλάσσουμε και την κυριαρχία των κρατών μελών, ενώ ταυτόχρονα μπορούμε και να προχωρήσουμε. Μπορεί μερικοί όμως να ε, που μήπως αυτές οι αυτοεξαιρέσεις θα καταστρέψει την ε, πολιτική οικονομία που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Ε, και θα πρέπει να δούμε πώς θα εξυπηρετήσουμε τις χώρες που θέλουν να αυτοεξαιρεθούν, όπως η Ιρλανδία με τον εταιρικό φόρο, για παράδειγμα. Θα μπορούσε να γίνει και αυτό, αλλά δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε αυτοεξαιρέσεις που θα καταστρέφουν την, την ένωση των πολιτικών που θέλουμε να φτιάξουμε με αυτή την υπερπλειοψηφία. Επίσης έχουμε τις διάφορες κατηγορίες χωρών πρέιν, πόστιν, πιθανά μέλη και τι γίνεται με τη δημοκρατική αποτελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ίσως πρέπει να δώσουμε φωνή και ψήφο στου, στους τομείς πολιτικών στους οποίους συμμετέχουν. Ε, Ελβετία για παράδειγμα, Νορβηγία αλλά και Τουρκία και κατά πάσα πιθανότητα και το Ηνωμένο Βασίλειο αν τελικά ε, το έγγραφο του Άντριου Ντάφ είναι προφητικό για το τι θα συμβεί με το Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά πρέπει να γίνει και μια επανισορρόπηση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Ο Ματίας Κούμα μας μίλησε για το θέμα αυτό, αλλά με την κρίση του ευρώ υπάρχει ε, πρόβλημα με υπερβολική τεχνοκρατία. Ε, γιατί κάτι τέτοιο θα επηρεάσει και το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή. Σε ό,τι αφορά την νομιμοποίηση το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Εκεί οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων πολύ συχνά υπενθυμίζουν και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι είναι οι πιο νομιμοποιημένοι γιατί αυτοί προσωπούν του Ευρωπαίου πολίτε. Αν όμω δούμε τα παζαρέματα που γίνονται διακυβερνατικά, εκεί που υπάρχει η νομιμοποίηση, όταν τα πιο ισχυρά κράτη είναι αυτά που πρωτοστατούν και καθορίζουν το θεματολόγιο. Ονόματα δεν λέμε. Πέραν τούτου, ε, σε ό,τι αφορά το, το διακυβερνητικό επίπεδο, έχουμε όλο και, ενίσχυση, όλο και μεγαλύτερη ενίσχυση αυτού του διακυβερνητικού επίπεδου, ιδιαίτερα στην κρίση του ευρώ. Οπότε καταστρέφουμε την κοινοτική μέθοδο, την υπονομεύουμε και παραγκονίζουμε ουσιαστικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τι χρειάζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλει να συμμετέχει πλήρως στη συζήτηση για την κρίση του ευρώ και της ευρωζώνης, ε, να μιλάει με την ευρωπαϊκή φωνή, να συμμετέχει το Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο στη συζήτηση για όλες τις πολιτικές. Βέβαια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρειάζεται και τη δική του πολιτική νομιμοποίηση. Μεγαλύτερη αντιπροσωπευτική ε, νομιμοποίηση. Και είπαν ε, οι κύριοι Κούμ και Μαντζέλα ότι αν στις Ευρωεκλογές του 2014 έχουμε ένα, και την υποψηφιότητα του Πρόεδρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προεκλογική διαδικασία θα προκαλέσει κάποιε συζητήσει ε, και για τι πολιτικέ στα κράτη-μέλη. Αυτό βέβαια θα αποτελέσει την απαρχή για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Πολύ πιθανόν. Αλλά αυτέ οι πορείε είναι πολύ χρονοβόρε. Για παράδειγμα, χρειάστηκαν 100 χρόνια για να αναπτυχθούν τα πολιτικά κόμματα ε, στι Ηνωμένε Πολιτείε. Ελπίζουμε να είναι πιο γρήγορη στι εξελίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Είπαμε προηγουμένως θα πρέπει να απεθνικοποιήσουμε τη διαδικασία αυτή. Ίσως όμως για να φτιάξουμε ε, πανευρωπαϊκά κόμματα, ίσως πρώτα θα πρέπει να επανέλθουμε σε μια εθνικοποίηση. Δεν μιλάω τώρα για τον πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά για του υπόλοιπου επιτρόπου. Γιατί να μην είναι οι επικεφαλεί των εθνικών ψηφοδελτίων. Οπότε θα έχουμε σοβαρέ ε, προσωπικότητε που θα είναι οι επικεφαλεί των ψηφοδελτίων και όποιο και αν εκλεγεί, όποιο και βρίσκεται στο συνασπισμό, ένα από τα μέλη του Εθνικού Κόμματο, που είναι και επικεφαλή του ψηφοδελτίου, θα φτάσει στη θέση του επιτρόπου. Βέβαια, το μόνο πρόβλημα με αυτό είναι τι θα συμβεί αν έχουμε συνέχιση της αποχής από τις ευρωεκλογέ. Θα υπάρξει πρόβλημα. Ή αν οι επίτροποι δεν, θεωρήσουν την υπουργή μιας κυβέρνησης, άσχετα από τις εκλογικές περιφέρειες, αλλά ε, κάτι αντίστοιχο σαν τους γερουσιαστές της, ε, των Ηνωμένων Πολιτειών. Ή να υπάρξει μια πολιτικοποίηση και αντιπαράθεση βορρά και νότου. Ή να έχουμε μια πόλωση προς τα άκρα. Αυτό μπορεί να συμβεί αν έχουμε μεγάλο ποσοστό αποχής η πολιτικοποίηση είναι ένας κίνδυνος πανταχού παρών. Το είδαμε, τον είδαμε και σε εθνικό επίπεδο. Γιατί μερικές φορές αυξάνεται η συμμετοχή με στις εθνικές εκλογές. Αλλά με τέτοια πολιτικοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο η κίνδυνη είναι μεγαλύτερη. Τώρα, γιατί έχει νόημα να γίνει κάτι τέτοιο παρά τους κινδύνους. Υπάρχει και μια άλλη πτυχή που σχετίζεται με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα έχει μεγαλύτερη πολιτική νομοποίηση ε, αντιπροσωπευτική, αντιπροσωπευτικότητας, γιατί θα έχει εκλεγεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί ε, στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μεγαλύτερη πολιτική και διοικητική ευχέρεια και ελαστικότητα κατά την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, για παράδειγμα. Γιατί ένα από τα προβλήματα, μερικά από τα προβλήματα που έχουμε σήμερα είναι το ότι η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, σε μερικού τομεί είναι λίγο κάτι παραπάνω από γραμματεία ουσιαστικά, εξαιτία τη αυτόματη εφαρμογή των κανόνων που επιβάλλουν. Υπάρχει αυτοματισμό στην εφαρμογή των ρόλων και στους αριθμούς. Ενώ αν έχουμε έναν εκλεγμένο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα έχουμε μια ουσιαστική, σοβαρή διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο. Και τώρα φτάνω στο θέμα της πολυεπίπεδης ε, διακυβέρνησης σε μια διαφοροποιημένη πολιτική οικονομία. Για να πραγματοποιήσουμε αυτή τη διακυβέρνηση και να είναι λειτουργική η οικονομία θα πρέπει να περάσουμε αυτό το σημερινό αυτοματισμό και την τεχνοκρατία τη σημερινή σε μια γνήσια ουσιαστική διακυβέρνηση. Τι σημαίνει όμως αυτό. Τώρα να εφαρμόσουμε μία λύση για όλους ε, δεν πρόκειται να λειτουργήσει. Ή να είναι οι, κυβέρ... κανόνες υποκατάστατο της διακυβέρνησης. Ούτε και αυτό μπορεί να είναι αποτελεσματικό γιατί δεν θα έχουμε συμφωνία για τις λεπτομέρειες. Το πρόβλημα τους ε, κανόνες είναι ότι οι λύσεις για το βορρά δεν ε, λειτουργούν στο νότο ή στην Ανατολή. Ιδιαίτερα θέλουμε να ε, ανατάξουμε την κατάσταση, να ε, προχωρήσουμε σε μια ανάκαμψη της οικονομίας και να προωθήσουμε την οικονομική ανάπτυξη. Υπάρχουν πολλές διαφορές, υπάρχουν διαφορετικές μορφές καπιταλισμού, διαφορετικά μοντέλα αναπτυξιακά στις διάφορες χώρες. Το πρόβλημα που έχουμε σήμερα είναι ότι γίνονται πολύ λόγο για τα αντικίνητρα, για τα φόβητρα μάλλον, για τα ραβδιά, αλλά δεν έχουμε καρότα, δεν έχουμε ενάψματα. Αν είχε όμω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεγαλύτερη πολιτική νομοποίηση και μεγαλύτερη ελαστικότητα, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Πώ θα ορίσουμε το έλλειμμα, για παράδειγμα, για τι χώρε στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Αν αφήναμε ε, αν δίναμε περισσότερες, ε, αφαιρώνουμε περισσότερες επενδύσεις ε, σε αναπτυξιακά προγράμματα, σε παιδεία και αν είχαμε ε, μεγαλύτερη νομοποίηση στις εκλογές και μεγαλύτερη πλειοψηφία και για την Επιτροπή θα μπορούσε, να το, θα μπορούσε να το κάνει. Να πούμε υπάρχει μια προοδευτική πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οπότε μπορούμε να ε, προωθήσουμε προοδευτικές πολιτικές. Αν είναι συντηρητική η πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθετούμε περισσότερο συντηρητικές πολιτικές. Πάντως έχουμε πολιτικοποιημένη ε, κατεύθυνση της πολιτικής, αλλά τουλάχιστον έχουμε μια μετάβαση από την τεχνοτροπία σε πιο πολιτικούς ε, νεοφιλελεύθερους κανόνες. Γιατί ούτως ή άλλως σήμερα είχαμε κανόνες που δεν ε, απέδωσαν, αλλά προβάλλονται σαν να είναι οι μοναδικοί κανόνες που είναι τεχνοκρατικοί και δεν είναι πολιτικοί. Στην ουσία όμως είναι και πολιτικοί και αυτό το γνωρίζει ο κόσμος. Γιατί να μην είμαστε λοιπόν πιο σαφείς, πιο ε, ξεκάθαροι με αυτά και να προχωρήσουμε και λίγο παραπέρα. Τώρα, ενισχυμένη συνεργασία. Σίγουρα η ενισχυμένη συνεργασία είναι αποτελεσματικό τρόπο. Ίσως θα πρέπει να τη χαλαρώσουμε κάπως και την ενισχυμένη συνεργασία. Ίσως α, ε, για λιγότερες χώρες Αυτές είναι οι ιδέες που προτείνω, μερικές μπορεί να λειτουργήσουν, άλλες όχι. Γιατί να μην έχουμε λοιπόν νέες ζώνες ενισχυμένης συνεργασίας, για παράδειγμα ενισχυμένες ζώνες κινητικότητας ε, του εργατικού δυναμικού και μια ολοκληρωμένη ε, αγορά εργασίας ε, με διάφορες μορφές ρύθμισης. Γιατί αν θέλουμε ε, πιο ε, ολοκληρωμένη εσωτερική αγορά και πιο βαθιά. Και μιλούμε και για κάποιες πτυχές της κοινωνικής πολιτικής, ε, αγοράς εργασίας, ακράτους πρόνοιας. Μπορούμε να το κάνουμε μόνο με ζώνες ενισχυμένης συνεργασίας, γιατί όχι και ζώνες κοινοφελών υπηρεσιών, υπηρεσίες υγείας, συμφωνίες ε, διασυνοριακής κινητικότητας, οι ζώνες μετανάστευσης, όπου χώρες με παρόμοιες ανάγκες θα αναρμονίζουν τις μεταναστευτικές τους πολιτικές. Υπάρχουν τέτοιες ε, λύσεις. Βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ε, ξανατονώσει την ευρωπαϊκή οικονομία, τη μεγαλύτερη ανάγκη για τους Ευρωπαίους πολίτες. Άρα ακούσαμε ε, την πρόταση για τα ομόλογα έργου. Σε τι φάση βρίσκονται. Θα ήταν χρήσιμα για επενδυτικά προγράμματα και σχέδια αυτά τα ομόλογα έργου. Για το σιδηροδρομικό δίκτυο, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ε, για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα ή για νέες ανανεωμένες βιομηχανικές ζώνες. για διάφορες αναπτυξιακές συνεργασίες ή τι γίνεται με τα διαρθρωτικά ταμεία. Και αυτά θα πρέπει να μεταρρυθμιστούν για να είναι πιο λειτουργικά, να είναι πιο ε, εύκολα προσπελάσιμα. Και υπάρχει και ένα έγγραφο για το θέμα αυτό. Γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε το χρησιμοποιητό τμήμα των διαρθρωτικών ταμείων για μόχλευση των επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Η αναθεώρηση της κοινή γεωρικής πολιτικής. Για πόσο καιρό μιλάτε για τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωρικής πολιτικής. Γιατί λοιπόν ε, να μην ε, προσθεθεί και στην ΚΑΠ ένας ε, φόρος για τους μεγαλοπτηματίες, για τους εκατομμυρίουχους ή ένα ασφαλιστικό ταμείο για, την, για τους ανέργους. Θα μπορούσαν τα διαρθρωτικά κονδύλια να αφιερωθούν και σε αυτούς τους σκοπούς. Βέβαια φυσικά κάτι τέτοιο απαιτεί ένα μεγαλύτερο κοινοτικό προϋπολογισμό, ενίσχυση του κοινοτικού προϋπολογισμού. Το πρόβλημα βέβαια είναι ότι αν πούμε στα κράτη-μέλη δώστε μας περισσότερα χρήματα, καταστροφή. Χρειαζόμαστε νέες πηγές εσόδων και αυτό το συζητήσαμε, τουλάχιστον το συζητάμε ακόμη, φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Γιατί όχι μέσω ενισχυμένη συνεργασίας μεταξύ ομάδων χωρών. Ήδη ασυνοριακό ε, φόρος ε, χρηματοπιστωτικών ε, συναλλαγών για αγαθά και υπηρεσίε για να αποφευθούν κάποια αρνητικά αποτελέσματα της ενίας αγοράς και να διορθωθούν κάποια περιβαλλοντικά προβλήματα. Ή φόρος αλληλεγγύης, για παράδειγμα, στους Ευρωπαίους πολίτες, για να, διαμορφώσουμε, για να ενισχύσουμε την αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών, για να μην φαίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο ε, για μια ένωση της μεταφοράς, όπου ένα τμήμα της Ευρώπης θα πληρώνει για την υπόλοιπη. Βέβαια, μερικοί θα πούν όχι στο φόρο αλληλεγγύης θα μπορούσε να είναι προαιρετικό για του πολίτε τη Μεγάλη Βρετανία, για να μην έχουμε πολλέ εταιρείε. Όχι, πλάκα κάνω. Εν πάση περιπτώσει, εγκατακλείδη. Με όλα αυτά τα νέα έσοδα και τι ευθύνε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη, οι πολίτε θα περιμένουν μεγαλύτερη πρόσβαση στη διαδικασία λήψεων αποφάσεων και φυσικά μεγαλύτερες ε, εγγυήσει για, για δημοσιονομική ε, πειθαρχία. Για όλα αυτά όμως χρειαζόμαστε βαθύτερη πολιτική ολοκλήρωση. Οπότε ε, εκλογή του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι η απαρχή για τη μεγαλύτερη δημοκρατική νομοποίηση και με συμμετοχή όλων των κοινοτήτων. Έτσι νομιμοποιείται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει τη γενική επίβλεψη για τις κοινοτικές πολιτικές. Φυσικά χρειάζεται και ε, καινοτόμο ηγετικό ρόλο του Συμβουλίου. Καλύτερη επικοινωνία προ το κοινό, που θα εξηγεί στο κοινό τι σημαίνει, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια είναι η, η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Χρειαζόμαστε συνεχή επικοινωνία με το κοινό, να εξηγούμε συνέχεια στους πολίτες τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιες είναι οι κοινοτικές πολιτικές θα πρέπει στην επικοινωνία αυτή να περιλάβουμε την αλληλεγγύη και την ευημερία, αντικαθιστώντας την ειρήνη και την ευημερία, ή ένα νέο ε, κοινωνικό νέο φιλελεύθερο μοντέλο, σε αντικατάσταση του νέου φιλελεύθερου μοντέλου. Γιατί μιλάμε για, την, για τις λύσεις της πολιτικής οικονομίας, μιλούμε για τους απότερους σκοπούς Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους ε, μεγάλους σκοπούς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως σε μια πολιτική οικονομία πολιτικής ε, ε, διαφοροποιημένη ολοκλήρωσης, φυσικά χρειαζόμαστε και μια πολύ πιο ενισχυμένη δημοκρατία. Νομίζω ότι αυτά είναι τα θέματα που μας απασχόλησαν περισσότερο σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε καθηγήτρια. Θα δώσω μέσα στο λόγο στον κύριο Γιάν Μπέκ, που είναι καθηγητής στη London School of Economics και κάνει έρευνα για διάφορα σημεία και στοιχεία της οικονομικής πολιτικής ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ε, επίσης ε, είναι διευθύνων ε, του Journal of Common Market Studies και ήταν και σύμβουλος της Βουλής των Λόρδων σε αντίστοιχα θέματα. Παρακαλώ. Α, έχετε έρθει ήδη στο Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν μπορώ να αντισταθώ στον πειρασμό να αρχίσω με μια πολύ μικρή ιστορία για κάτι που συνέβη την περασμένη Κυριακή. Θα γνωρίζετε ότι στο γκολφ ήταν το Ryder Cup. Και ε, οι περισσότεροι που παίζουν ε, στο γκολφ είναι ευρωσκεπτικιστέ στην Αγγλία και ε, παρόλα αυτά υποστήριζαν την ευρωπαϊκή ομάδα που τελικά νίκησε τη Ryder Cup. Ε, για να δείτε πώς λειτουργούν οι ευρωσκεπτικιστές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, θα ήθελα να μιλήσω για τη δημοσιονομική διάσταση. Ε, είναι ακριβώς το ακαθόδες θέμα. Πρόκειται εδώ ακριβώς για ε, τα χρήματα και για το πώς θα πιστούν οι πολίτες. Στην αλληλεγγύη και σε αυτό το εγχείρημα θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε γιατί έχουμε καν μηχανισμούς αλληλεγγύης. Και η πρώτη απάντηση είναι για την αναδιανομή. Χρειαζόμαστε να αναδιανέμουμε μέσω της αλληλεγγύης ε, τον πλούτο από το μία κοινωνική ομάδα σε άλλη. Αυτό μπορεί να γίνει αυτόματα με μηχανισμούς φορολογικούς και επιδομάτων που είναι μεταφορές ε, πιστώσεων μεταξύ ε, ατόμων ή μπορεί να υπάρξει μια ροή κεφαλαίων από μια κυβέρνηση, από ένα οργανισμό που αποφασίζει ότι ορισμένες κοινωνικές ομάδες θα ευνοούνται από αυτές τις μεταφορές. Ε, το άλλο είδος είναι με τη φορολογία ε, και τα προοδευτικά φορολογικά συστήματα προχωρούν όσο αναδιανέμουν από τους ε, πλούσιους τους στοχούς βασικά. Και ε, στο ευρωπαϊκό πλαίσιο θα πρέπει να σκεφτόμαστε πάρα πολύ προσεκτικά το θέμα των δανείων και πώς αυτά συμφωνούνται. Γιατί για να κερδίσει κάποιος ένα πλεονέκτημα από ένα συγκεκριμένο κράτος ή μια επικράτεια του είναι να τους δίνουμε δάνεια με πολύ πιο ευνοϊκούς όρους από όσο θα μπορούσαν μόνο τους να πάρουν. Και αυτό έχει και ένα δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Και παρόλη την ε, ροή κεφαλαίων και στην Ευρώπη τι έχουμε σήμερα. Πάρα πολύ ε, λίγο, πολύ λίγες διασυνοριακές εκταμιεύσεις πέραν ε, των ε, δωρεών ας πούμε από το Ταμείο Συνοχής ε, και το Ταμείο της Γεωργίας για την κοινή γεωργική πολιτική. Αλλά σε καμία περίπτωση αυτό δεν είναι διακρατικές ε, ε, εκροές. Σε αντίθεση με αυτό που σημαίνει στο εσωτερικό μιας χώρας που είναι πολύ διαφορετικού χαρακτήρα. Και ένα από τα προβλήματα της Ευρωζώνης είναι ότι δεν έχουμε καμία δυνατότητα σταθεροποίησης από τα πάνω προς τα κάτω εκτός του διάβλου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τώρα θα μου πείτε τι δουλειά έχει εδώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μα δίνει ρευστότητα με πάρα πολύ ευνοϊκού όρου και έτσι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ουσιαστικά δρά ω δημοσιονομική αρχή ε, και φορολογική. Δίνει πάρα πολύ ε, φτηνά δάνεια για να μπορούν τα κράτη-μέλη να χρηματοδοτούνται. Αυτό λοιπόν είναι το πλαίσιο του τι κάνουμε και τι δεν έχουμε. Ε, τι σχεδιάζει ένα πολυεπίπεδο σύστημα. Είναι δυτή η οικονομική λογική που κρύβεται από πίσω. Σε οποιαδήποτε νομισματική ένωση κάπου χρειάζεται στο σύστημα μια δυνατότητα σταθεροποίησης. Αυτό τι σημαίνει. Να προσπαθήσουμε να βεβαιωθούμε ότι ε, πηγαίνουν τα χρήματα στις οικονομίες που υφίστανται και πλήττονται από ασύμετρους ε, κραδασμού ε, σοκ. Ακούσαμε προηγουμένω για τον Τέξα τι έγινε. Ότι από πάνω προς τα κάτω η ροή των ε, πόρων ε, είναι και προς το συμφέρον ε, εκείνου που λαμβάνει τους πόρους αλλά και εκείνου που δίνει. Επίσης υπάρχει το θέμα της ισότητας για να υπάρχει μια σχετική ευημερία σε διάφορα μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένουμε οι πιο πλούσιες περιφέρειες σε ένα κράτος, μέλος η Βάδη Βιρτεμβέργη ας πούμε, προς το Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία ή από χώρα σε χώρα, η Σουηδία προς τη Ρουμανία, για λόγους ισότητας. Βέβαια, όταν έχει κάποιος ένα μεγάλο πρόβλημα, μεγάλη διαφορά ε, και μπορεί να σπάσει ε, ο, ο κύκλος αυτός της ανάπτυξης, αλλά υπάρχει και η προσωπική αλληλεγγύη και ισότητα ε, στη δημοσιονομική αλληλεγγύη και δεν μπορούμε να το ξεχνούμε αυτό είναι και η διαπροσωπική σχέση των ανθρώπων ιδιαίτερα όταν έχουν αντίστοιχο εισόδημα. Ποιο είναι το πρόβλημα με το Ταμείο Συνοχής αλλά το πρόβλημα είναι ότι η φτωχοί των πλουσίων χωρών χρηματοδοτούν τους πλουσίους των φτωχών χωρών, ανάλογα με το πώς χρησιμοποιούνται τα κράτη. Τώρα έχουμε εδώ και πολλούς ε, δικηγόρους ε, στην αίθουσα. Όταν έχουμε συνταγματικά εμπόδια δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα σε μια ε, συνθήκη, γι' αυτό έχουμε και αυτά τα εμπόδια. Περί τίνος πρόκειται λοιπόν, θα πρέπει να συμφιλιώσουμε τις διάφορες αντιστάσεις σε τις διάφορες ε, διαμάχες και τριβές για να παραμείνει ε, αυτή η ε, ισορροπία. Έχει πολύ σοφούς η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Μάρκ Τουέιν είπε ότι όποιος έχει μια νέα ιδέα θεωρείται τρελός μέχρι να πετύχει η ιδέα του. Και αυτό είναι το leitmotiv που κρύβεται πίσω από την οποιαδήποτε δράση. Να σκεφτούμε πέρα από τα θεσμικά πλαίσια, από τα εφικτά πολιτικά δεδομένα που έχουμε τώρα, να βγούμε παραπέρα, <laughs> να κάνουμε προτάσεις μέχρι και 23 διαφορετικές προτάσεις. Λοιπόν, ας βγω από το πλαίσιο. Ε, ορισμένες από τις ιδέες ε, είναι αμυγός δημόσια οικονομικά. Θα μπορούσαμε να έχουμε ένα σύστημα εκταμιεύσεων μονίμων νεκρών με κάποιο τρόπο και αυτό θα μπορούσε να είναι με ε, διακυβερνητική συνεργασία, δηλαδή το ευρωπαϊκό επίπεδο θα έχει περισσότερους πόρους για να μπορεί να τους χειρίζεται και να τους χρησιμοποιεί έτσι ώστε να εξισορροπεί τη ζήτηση από διάφορα μέρη της Ένωσης. Ποιο είναι εδώ το πρόβλημα, όπως είπε η Βίβιαν. Αν δεν μπορεί να αυξηθεί το εισόδημα, ε, μάλλον να έχει πόρους η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό. Και δεν μπορεί να υπάρχει φορολόγηση χωρί εκπροσώπηση. το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακριβώ το αντίθετο. Εκπροσώπηση χωρί φορολόγηση. Δεν υπάρχει δυνατότητα επιβολή φόρων σε κοινοτικό επίπεδο. Μόνο τα κράτη-μέλη μπορούν να το κάνουν. Το άλλο είναι αυτό που λένε στα γερμανικά Finanzausgleich, που είναι ο συμψηφισμό δηλαδή οριζόντιο, με όλε τι δυσκολίε που έκοσαμε στη Γερμανία. Μια οριζόντια μεταφορά πιστώσεων μεταξύ των ομόσπονδων κρατηδίων ή μεταξύ των κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δούμε το, ευρωπαϊκό, το γερμανικό συγγνώμη, παράδειγμα, δεν είναι πάρα πολύ αισιόδοξη η κατάσταση γιατί ε, πυροδοτεί ε, πιο έντονο ανταγωνισμό. Αλλά αυτές είναι οι δύο δυνατότητες ανάλυσης που έχουμε. Και στις δύο περιπτώσεις φαίνεται ε, ότι το κίνητρο είναι η αναδιανομή. Δηλαδή θέλουμε να μεταφέρουμε τα χρήματα από, από τον πλούσιο στο λιγότερο πλούσιο. Ε, αυτό είναι το θέμα με τη μεταφορά πιστώσεων. Ε, η αλληλεγγύη μπορεί να επιτευχθεί και με διάφορα προσωρινά μέτρα. Και τα έχουν συζητήσει οι οικονομολόγοι όλα αυτά τα χρόνια. Ας πούμε, το Ταμείο Ενεργείας που υπάρχει στη Φιλανδία, ότι σε καλούς καιρούς ε, ε, εισφέρεις και τα παίρνεις πίσω σε χαλεπούς καιρούς. Ε, βέβαια, θα, πρέπει να είναι ένα είδος ασφάλισης. Ε, πληρώνεις και όταν ε, βγεις στην ανεργία ε, παίρνεις ε, τα χρήματα, αλλά ε, το συνολικό υπόλοιπο είναι μηδέν. Άρα είναι και αυτό προσωρινό μέτρο, μεταβατικό. Η συνθήκη προβλέπει ορισμένες χώρες να τραβούν εκτάκτως χρήματα όταν τα χρειάζονται και να τα επιστρέφουν όταν δεν τα χρειάζονται. Αυτό τι σημαίνει ε, ισχυρούς όρους και προϋποθέσεις. Και εδώ μια λέξη κλειδί για να καταλάβουμε πώς μπορεί να λειτουργήσει η αλληλεγγύη είναι η αιρεσιμότητα. Δεν εννοώ με τον τρόπο που γίνεται σήμερα και αντιστέκεται η Ισπανική κυβέρνηση ή ε, ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει ε, ε, αντιδρούν οι Πορτογάλοι, οι Ιρλανδοί, οι Έλληνες. Έχει πολύ μεγαλύτερη σχέση εδώ και συνοχή με την αλληλεγγύη, γιατί η αλληλεγγύη σημαίνει έχεις πρόβλημα, θέλουμε να σε βοηθήσουμε, όχι είσαι φτωχός και θέλουμε να σε βοηθήσουμε. Είναι διαφορετική προσέγγιση, ηθικά τουλάχιστον. Δηλαδή είναι μια ατυχία, ε, όχι κάτι ε, μακροπρόθεσμο και διαφορές επίπεδα ευημερίας. Ε, ένας άλλος τρόπος να το εξετάσουμε είναι πώς μπορούν τα δημόσια οικονομικά να υποστηρίξουν τις χρηματορροές. Ιδιαίτερα να είναι πιο εύκολο να εκχωρούνται δάνεια ε, με βάση την αλληλεγγύη. Η απάντηση είναι ότι υπάρχει το μηχανισμό σταθερότητα στο άρθρο 122 και 143 για προβλήματα ισοζυγίου πληρωμών ή για έκτακτε περιστάσει. Αυτά υπάρχουν στη συνθήκη και θα μπορούσαν να επεκταθούν για να είναι αυτέ οι ροέ πιο αποτελεσματικές και με μόχλευση για να υπάρχει δυνατότητα ε, μεγαλύτερης δανειοδότησης και δανειοληψίας. Να είναι πιο εύκολο λοιπόν και πιο φτηνό να δανείζεται μια χώρα. Όπω μπορεί να γίνει μέσω αυτού του διάβλου. Όπως γνωρίζουμε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατέληξε σε αυτό που, το περίφημο που είπε ο Ζαν Κλώτρισε σε ε, μη συμβατικά μέτρα. Τι είναι αυτό, χρηματοδότηση του κόστους. Αλλά τι κάνουν πραγματικά. Στρεβλώνουν και ε, την ε, εντολή από τη συνθήκη, ε, την επεκτείνουν όσο μπορούν και την ταλαιπωρούν μέχρι του βαθμού που αντέχει να είναι ακόμα νόμιμη. Γιατί στις μεταφορές πιστώσεων από τους αποταμιευτές σε εκείνους που δανείζονται και μάλιστα πολλέ φορέ ε, είναι από χώρε που έχουν υπερβολική τάση στην αποταμίευση. Ε, εδώ όμω υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει Ευρωπαίος φορολογούμενος. Και απουσία του Ευρωπαίου φορολογουμένου τέτοιε ε, ροέ κονδυλίων είναι πάρα πολύ δύσκολο να δικαιολογούνται και να εξηγούνται σε εκλογικά σώματα. Γιατί οι φορολογούμενοι είναι ένα εθνικό εκλογικό σώμα. Ποιε είναι οι διαφοροποιημένε τώρα επιλογέ, Τι εννοώ αυτό που έχουν να επιλέξουν ορισμένα κράτη-μέλη, ομάδες κρατών μελών. Εδώ το πιο προφανές θα ήταν να πούμε γιατί δεν μπορεί η Ευρωζώνη να δημιουργήσει το δικό της προϋπολογισμό, ξεχωριστό από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, με τρόπο που να υπάρχει δυνατότητα να αντιμετωπίζει ειδικά προβλήματα σταθεροποίηση, μπορεί να είναι αυτό διάσωση, μπορεί να είναι ακόμα και ένα είδος ε, αναδιανομής ή αναζωγόνησης της μεγέθυνσης της οικονομίας. Η σταθεροποίηση είναι εύκολη. Αυτό τώρα που χρειάζεται είναι να δοθεί σάρκα και οστά στην ε, ε, Δημοσιονομική Ένωση. Πολύ διατυμπανίζεται αυτό, αλλά πολύ λίγο ορίζεται. Είναι τρία επίπεδα. Ε, είναι Ένωση Κανόνων, αυτό θέλουν οι Γερμανοί. Το δεύτερο είναι η Ένωση Ευρωμολόγων, αυτό που θέλουν οι Γάλλοι δηλαδή, και συνένωση του χρέους. Και το τρίτο είναι η Ένωση ε, των Μεταφορών Πιστώσεων. Και ε, αυτό το θέλουν όσοι λαμβάνουν τα χρήματα και δεν λέω ονόματα εδώ. Αλλά δεν υπάρχει ακόμα ορισμός για τη Δημοσιονομική Ένωση, αλλά με καθησύχασε αυτό που είπε ο Μπρούνο Ντεβίτ και ο Ζαν που δεν φημίζεται για την υποστήριξη τέτοιων ιδεών κατά τα άλλα. Από εκεί και πέρα τι μπορούμε να κάνουμε. Ενισχυμένη συνεργασία ε, ως ένα νέο μέσο για την επιβολή νέων φόρων, ιδιαίτερα το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Ενδεχομένως να είναι ένας τρόπος να δημιουργηθεί ιδίως πόρος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εγώ είμαι απεσιόδοξο σχετικά με αυτό. Δεν μπορώ να φανταστώ να συμφωνούν οι Βρετανοί και αφού είναι ομοφωνία, αμφιβάλλον θα μπορέσουν οι άλλοι να το περάσουν. Πάντως υπάρχει δυνατότητα να έρθει νέος φόρος με ενισχυμένη συνεργασία και στο μέλλον να είναι ένας τρόπος να βρεθούν χρήματα λιγότερο για το προϋπολογισμό της Ένωσης αλλά για άλλου είδους, ας πούμε ένα προϋπολογισμό Ευρωζώνης. Τρίτη προσέγγιση είναι ποιο θα συμφωνήσει να συνενωθεί το χρέος, ε, υπάρχει κοινή ευθύνη. Ε, παρόλες ε, ενάρετες και αξιέπαινες προτάσεις τα ευρωμόλογα, να τα ονομάσει ομόλογα έργο Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γερμανία δεν είναι πρόθυμη το δεχτεί. Είναι ένας τρόπος να μειωθεί ε, ε, το κόστος ε, για τις χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Τελικά σχόλια, καταληκτικά. Αν θέλουμε πραγματικά κάτι που θα ονομάσουμε πολιτική δημοσιονομική ένωση, θα πρέπει να κάνουμε και κάποιες θυσίες. Να καταλάβουμε ότι το status quo είναι απαράδεκτο αν θέλουμε να προχωρήσουμε σε αυτές τις νέες δομές. Χρειαζόμαστε ιδέες για τους μηχανισμούς. Και μπορεί αυτό να έχει επιπτώσει και τα θεσμικά όργανα. Γιατί, α πούμε, όταν έχουμε ευρωομόλογα, είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό χωρί ένα Ευρωπαϊκό Υπουργείο Οικονομικών. Κάποιο θα πρέπει να τα χειρίζεται. De facto υπάρχει αυτό ε, που είναι ε, το EFSF ε, είναι ξεχωριστό μηχανισμό υπό τον κύριο Κλάου Ρέγκλινγκ, πολύ περιορισμένο για Υπουργείο Οικονομικό, αλλά είναι ένα πρωτόλιο. Επίση, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν κίνδυνοι αν πάρουμε αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει κίνδυνο να διχαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σε κράτη-μέλη τη Ευρωζώνης και με τους υπόλοιπου 27 ή ακόμα και διάφοροι σχηματισμοί που φαίνονται ε, σε αυτά που είπε ο Βέσελ το πρωί, 25 που συμμετέχουν στο Δημοσιονομικό Σύμφωνο και άλλοι αριθμοί για άλλες πολιτικές, για άλλες προσεγγίσεις που έχουν να κάνουν με τη συνένωση του χρέους. Όλα αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε μεγάλα προβλήματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τον ηθικό κίνδυνο. Δεν μπορούμε να γνωρίσουμε να παραγνωρίσουμε ότι κάποιες προτάσεις και για την Τραπεζική Ένωση θα δημιουργήσουν κάποιο παθητικό που πρέπει να αντιμετωπιστεί από τα κράτη-μέλη. Και αυτό μας οδηγεί και πάλι ε, στο θέμα της νομιμοποίησης. Τελικά ποιος θα εκπροσωπεί τους φορολογουμένους, έχοντας υπόψη ε, αυτό που είπα προηγουμένω, ότι δεν υφίσταται Ευρωπαίο φορολογούμενο, είναι εθνικό φορολογούμενο. Ποιο θα του εκπροσωπεί, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα Εθνικά Κοινοβούλια, κάποιο άλλο. Τώρα σα πω κάτι που είπε ο Μάρξ και συνοψίζει τις συζητήσεις που κάνουμε. Θα το διαβάσω και πάλι. Η πολιτική είναι ε, ε, η τέχνη να ψάχνεις για προβλήματα, να τα βρίσκεις παντού, να τα διαγνώσεις με λάθος τρόπο και να εφαρμόζεις τις λάθος λύσεις. Στο κομμουνιστικό μανιφέστο δεν θα το βρείτε ούτε στο κεφάλαιο γιατί δεν είναι του Καλ Μάρξ, είναι του Κράουτσο Μάρξ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά. Και τώρα θα ακούσουμε τον τελευταίο ομιλητή καθηγητή σε πολλά πανεπιστήμια. Αυτή τη στιγμή κατέχει την έδρα του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Humboldt του Βερολίνου. Ε, ελάτε, αν θέλετε, στην έδρα. Και είναι αυτή τη στιγμή εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου ε, του Διεθνούς και Συνταγματικού και βεβαίως θα μπορέσουμε να κάνουμε και κάποιες ερωτήσεις μετά ε, ναι, εργαστήκαμε το ή άλλως αρκετά σήμερα ε, οι συνάδελφοι που είναι εδώ μπορούν ίσως να προημαστούν για να κάνουν κάποιες ε, παρεμβάσεις Ευχαριστούμε. καθίστε όπου σας βολεύει. Ίγκολφ. Ούμπολτ είναι το πανεπιστήμιο, μάλιστα. Έχετε το λόγο λοιπόν. Ε, ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, για την ευκαιρία που μου δίνετε να βγάλω συμπεράσματα από μια πάρα πολύ συναρπαστική ημέρα και οπωσδήποτε δεν θα επαναλάβω αυτό το οποίο ακούστηκαν. Ξέρω ξεπερνώ τις δυνατότητες μου. Ξεπερνά τις δυνατότητες μου κάτι τέτοιο. Το θέμα λοιπόν το σημερινό για το μέλλον της ε, πολλαπλής διακυβέρνησης στην Ευρώπη έχει ένα νόημα διτό από ό,τι κατάλαβα. Το ένα είναι πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και το άλλο ε, είναι διακυβέρνηση πολλών ταχυτήτων. Νομίζω ότι αντιμετωπίσαμε και τις δύο πτυχές, θα έλεγα, σήμερα. Να ξεκινήσω με το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε όλοι σήμερα και το γιατί όλη αυτή η διαδικασία του να επανεξετάζουμε την Ευρώπη ξεκίνησε. Ξεκίνησε αυτό μια διέξοδο από την Ευρωκρίση. Όπως αντιλαμβάνομαι εγώ, πρέπει σήμερα να δούμε πώς ο μηχανισμός σταθερότητας και το δημοσιονομικό σύμφωνο θεωρήθηκαν αναγκαία μέσα έτσι ώστε προσωρινά τουλάχιστον να αντιμετωπίσουμε την κρίση. αλλά είναι σαφές πως υπάρχει μία ανάγκη να επαναπατριστούν αν θέλετε, να ενταχθούν αυτά τα μέσα στο θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης για να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα που είχαμε με το όχι της Μεγάλης Βρετανίας και της Τσεχίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από ό,τι φαίνεται δεν επηρεάστηκε από τα νέα αυτά μέσα, αλλά αντιθέτω, τα νέα αυτά μέσα προσφέρουν και ευκαιρίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να επεξεργαστεί πολιτικές και να ελέγξει κάποια, να κάποια πράγματα τα οποία δεν είχε τόσο εύκολα στο παρελθόν. Οπότε δεν ήταν απειλή αυτό στο, για το Κοινοβούλιο, αλλά μια ευκαιρία για να αποκτήσει έλεγχο σε που ήταν στα χέρια των κυβερνήσεων. Ένα άλλο ζήτημα είναι το άρθρο 125 μια διάταξη η οποία θα αποτελούσε εμπόδιο εάν δεν άλλαζε το άρθρο 136 και η παραγραφός 3 ε, καθώς θα δημιουργούσε προβλήματα για τον μηχανισμό σταθερότητας. Εγώ θα έλεγα ναι, υπάρχει μία αρκετά διαδεδομένη και κλασική άποψη πως η ρήτρα μη διάσωσης είναι εμπόδιο, αλλά θα έλεγα επίσης πως υπάρχουν και άλλες απόψεις που λένε πως η ρήτρα μη δεν ε, απαγορεύει την εθελοντική βοήθεια από το ένα κράτος μέλος στο άλλο ή θα αποκλεί κάποια δάνεια πίστοσης απλά αποκλεί την ευθύνη ενός κράτους μέλους για το χρέος τα προβλήματα μιας άλλης ή τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν αυτή την ευθύνη. Και αυτό είναι ένα μήνυμα που απευθύνεται στις χρηματαγορές, στις τράπεζες. Προσέχετε, δηλαδή, αν δανείζετε σε ένα κράτος μέλος, να είστε σίγουροι πως δεν θα σας εξοφλήσει άλλο κράτος μέλος ή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν Σημαίνει αυτό λοιπόν πως δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να βοηθήσει ένα κράτος κάποιο άλλο. Απλά επισημαίνω αυτή τη δεύτερη ερμηνεία γιατί μπορεί να τεθεί το ζήτημα ενώπιον του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου και ίσως και ενώπιον του ΔΕΚ και αν η απόψη είναι ομόφωνη πως ο μηχανισμός σταθερότητας είναι αντίθετος με το άρθρο 125 θα έχουμε πρόβλημα. Για το μακροπρόθεσμο πλαίσιο τώρα. Θεωρώ πως είναι αναγκαίο να ενσωματωθούν οι μηχανισμοί του Δημοσιονομικού Συμφώνου στο Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο και να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή δημοσιονομική και οικονομική πολιτική, κάτι το οποίο δεν σημαίνει πως θα αφαιρεθεί η αρμοδιότητα του προπολογισμού από τα κράτη-μέλη, αλλά σημαίνει πως βλέπουμε το ότι οι αποφάσεις του ενός κράτους μέλους μπορούν να επιδρούν στην ε, αυτονομία του προπολογισμού ενός άλλου κράτους μέλους. Και αυτό μας το δείχνει το παρελθόν. Εάν η Ελλάδα είχε άλλη δημοσιονομική πολιτική, ίσως να μην είχαμε τα προβλήματα που έχουμε σήμερα. Εάν η Γερμανία είχε άλλη δημοσιονομική πολιτική, μπορεί να μην είχαμε τα προβλήματα που έχουμε σήμερα στην Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα. Οπότε υπάρχει μια σχέση εδώ πέρα, μια αλληλεπίδραση και αυτό δεν έχει ληφθεί υπόψη και θεωρώ πως δεν έχει χαθεί η αυτονομία στο πλαίσιο της εθνικής κυριαρχίας του υπερβολισμού, αλλά ίσως έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα όπως αυτά που έχουμε σήμερα, η ευρωκρίση, ε, πολύ καλύτερα στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Οπότε και πάλι θα υπήρχε εθνική κυριαρχία ε, όσον αφορά τον προπολογισμό. Να έρθω τώρα στο δεύτερο ε, σημείο. Έχω πέντε από αυτά. Είναι το ζήτημα των κομματιών εκείνων που αφορούν τις οικονομικές και πολιτικές. Δηλαδή, εάν θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να χωριστεί και να πούμε πως εάν συζητάμε ζητήματα Ευρωζώνης, μόνο αυτό το κομμάτι του Κοινοβουλίου μπορεί να είναι παρόν στη συζήτηση. Ή, ή να πούμε Δευτέρα με Τετάρτη έχουμε τις γενικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Πέμπτη και Παρασκευή. Πέμπτη και Παρασκευή έχουμε μόνο τους ευρωβουλευτές των χωρών της Ευρωζώνης. Η εντύπωσή μου είναι πως ε, υπάρχει μια άσχημη αίσθηση για κάτι τέτοιο. Είναι αντίθετο με την ιδέα της ενότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήταν ένα κομμάτι του πολιτικού μεσιανισμού που ανέφερε ο Τζόζεφ Βάιλερ. Έχουμε μία Ευρωπαϊκή Ένωση και εδώ πέρα δεν έχουμε μία κοινότητα της μοίρα για πάντα, ας πούμε, όπως είναι ένα εθνικό κράτος, αλλά κάτι το οποίο πρέπει να ενώσει τους λαούς της Ευρώπης και το να διασπάσουμε τα θεσμικά όργανα σημαίνει κατακαιρματισμό και υπάρχει δυσκολία ε, όσον αφορά την εμπιστοσύνη στα θεσμικά όργανα εάν οι εντάσεις αυτές ε, γίνουν καθημερινός ε, διχασμός. Οπότε θεωρώ πως καλύτερο θα ήταν να βρούμε άλλες λύσεις. Οπότε κάποια πράγματα δεν νομίζω πως ε, χρειάζεται να γίνει τέτοιος διαχωρισμός για το κοινοβούλιο ή το δικαστήριο ε, να συζητήσουμε αν θα χρειαζόταν ας πούμε, αν θα ήταν χρήσιμο για την Κομισιόν. Εξάλλου, η Κομισιόν δεν είναι πρέσβη των κρατών μελών. Αντιθέτω, δεσμεύονται από τη συνθήκη ε, να εκφράσουν το ευρωπαϊκό συμφέρον. Οπότε γιατί μια ευρωπαϊκή ευρωζώνη να μην είναι προς το συμφέρον της Ένωσης στο σύνολό τη. Και οι ευρωβουλευτές εσείς δεν είστε πρέσβεις των χωρών σας. Είστε πρέσβεις, ε, εκπρόσωποι αν θέλετε, κάποιων περιοχών, ε, λαών αλλά δεν ε, εκπροσωπείται εθνικά ε, συμφέροντα αλλά έχετε μια εντολή να υπηρετείτε και το ευρωπαϊκό συμφέρον. Ακόμα και έτσι λοιπόν θα προτιμούσα πολλοί από του συμμετέχοντε να συμφωνούν με την άποψη αυτή πως δεν θα πρέπει δηλαδή να υπάρξει τέτοιο διαχωρισμός. Να έρθω τώρα στο τρίτο σημείο. νέε. αρμοδιότητε για την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αναφέρθηκε ήδη. Ευθύνη για δημοσιονομικές και οικονομικές πολιτικές και που θα συμπεριλαμβάνουν και μεγάλη αύξηση των πόρων του προϋπολογισμού θα ήταν το κάτι το επιθυμητό αυτό κατάλαβα εγώ τη συζήτηση. Δεν υπάρχουν πολλά λεφτά στο ευρωπαϊκό επίπεδο, ας πούμε πως τα διαρθρωτικά τα μία ή άλλα αποκτούν περισσότερους πόρους από όσους έχουν αυτή τη στιγμή και υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες υπάρχει, για απαιτείται ας πούμε κάποια επιδότηση για την ανάπτυξη και την ε, οικονομική δραστηριότητα σε κάποιο κράτος μέλος. Βεβαίως, εάν μεταφερθούν αυτές οι πολιτικές ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν κάποια όρια όπως ξέρετε τα οποία έχουν τεθεί και προσφάτως από το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο, αλλά να θυμάστε πως το δικαστήριο στην τελευταία του απόφαση αναφέρθηκε στην απόφαση του περί Μάστριχτ, όπου λέγεται πως ε, στην περίπτωση που η ασύμμετρη δομή της ΟΝΕ δεν ε, λειτουργεί, μπορεί να υπάρξει μεταρρύθμιση, κάτι το οποίο σημαίνει πως ε, υπάρχει περιθώριο ε, για αρμοδιότητες στο ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα των δημοσιονομικών και του προπολογισμού για να σωθεί το ευρώ, αλλά βεβαίως υπάρχουν όρια. Δεν μπορεί να αφαιρεθεί το δικαίωμα της γερμανικής βολής ή οποιοδήποτε άλλου κοινοβουλίου να έχει τον τελευταίο λόγο επί του προϋπολογισμού του. Αλλά οπωσδήποτε μπορούν να μπουν όρια, ένα πλαίσιο εντός του οποίου, ένα διάδρομο αν θέλετε, εντός του οποίου θα κινηθούν οι εθνικές πολιτικές για να υπάρχει μια οικονομική συνοχή εντός της Ένωσης προς όφελος ε, της επιβίωσης του ευρώ. Είμαι σίγουρος πως αυτό είναι δυνατόν. Όμως, αυτό θα αντικατοπτρίζει και την ε, επίδραση και τις σχέσεις ε, των εθνικών πολιτικών. Και πάλι, όπως είπα, δεν πρέπει να τον γνωρίσουμε μια απώλεια αρμοδιοτήτων. Κάτι άλλο, το επόμενο, αφορά την νομιμοποίηση και αφορά την εμπλοκή των εθνικών κοινοβουλίων που συζητήσαμε και από ό,τι καταλαβαίνω ε, και ερμηνεύω τη συζήτηση δεν ήθελε κανείς να δημιουργηθούν νέοι φορείς και θεσμικά όργανα εντός των οποίων τα εθνικά κοινοβούλια θα εκπροσωπούνται. Τα εθνικά κοινοβούλια κατά βάση υπάρχουν για να ελέγχουν και να νομοποιούν τις εθνικές πολιτικές. Αλλά όσο ισχύει πώς ο, η βασική πηγή της νομοποίησης της, ε, των ευρωπαϊκών πολιτικών όπως αναφέρεται και στο άρθρο 10 της συνθήκης ε, της Ένωσης είναι τα εθνικά κοινοβούλια αυτό το οποίο θα χρειαζόμασταν λοιπόν πολύ περισσότερο από νέα θεσμικά όργανα είναι ενημέρωση για την ευρωπαϊκή διάσταση και την ευρωπαϊκή λειτουργία και τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα των Εθνικών Κοινοβουλίων που δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή ως ε, δεν τίθεται ως συζήτημα και αν γίνει σαφές πως τα Εθνικά Κοινοβούλια έχουν ένα ρόλο να παίξουν μέσω του ελέγχου των κυβερνήσεων που είναι στο Συμβούλιο έχουν ρόλο λοιπόν στην ευρωπαϊκή πολιτική τότε η δυνατότητα του, των βουλευτών στα Εθνικά Κοινοβούλια η δυνατότητα συμμετοχής στην, σε ευρωπαϊκές συζητήσεις. Τότε αυτά τα ζητήματα θα ήταν ζήτημα στις εθνικές εκλογές, οι οποίες θα γίνονταν όλο και περισσότερο ευρωπαϊκές σε χαρακτήρα. Όπως ακριβώς ζητάμε και οι ευρωπαϊκές εκλογές να ε, είναι περισσότερο ευρωπαϊκές και όχι μόνο εθνικές σε χαρακτήρα. Με αυτή την εκπαίδευση λοιπόν των Εθνικών Κοινοβουλίων θα μπορούσαμε να αυξήσουμε και την νομοποίηση των εθνικών των ευρωπαϊκών πολιτικών, με συγχωρείτε από τους πολίτες. Ενισχυμένη λοιπόν δημοκρατική νομοποίηση. Η ανάλυση του Τζο Βάιλερ για τη δημοκρατία χωρίς το λαό και την έλλειψη Δήμου νομίζω ήταν ξεκάθαρη. Περιέγραψε το πώς έχει κατάσταση τώρα. Το ζήτημα είναι πώς οι ευρωπαϊκές εκλογές θα γίνουν εκλογές μιας πραγματικής πολιτικής επιλογής. Αναφέρθηκαν παραδείγματα. Κάθε ομάδα κόμμα, κάθε κόμμα, με συγχωρείτε, ορίζει έναν υποψήφιο για πρόεδρο της Κομισιόν Καλό θα ήταν αυτό γιατί θα υπήρχε έτσι και ένα πρόσωπο που θα διαλέγαμε στις εκλογές. Διαλέξουμε μεταξύ του κυρίου Σούλτς ας πούμε και κάποιο από το ΕΛΚ ας πούμε, δεν ξέρω, από την Ισπανία ή την Ιταλία. Καλό θα ήταν αυτό. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε κατά νου αυτή την ιδέα ότι επίτροποι στο μέλλον θα μπορούσαν να κατεβαίνουν σε κάποιες εθνικές λίστες για τις ευρωεκλογέ. Αλλά βεβαίω τα άτομα αυτά ε, είναι άτομα. Πρέπει να συνδυαστούν και με πολιτικά προγράμματα τα οποία δεν μπορεί να είναι μόνο στα χαρτιά αλλά να έχουν και όνομα οπότε δεν θα είναι μια ουδέτερη ε, διοικητική μηχανή όπως πιστεύουν μερικοί ακόμη και ο πρόεδρος ακόμη και να εκλέγεται με πολιτικό πρόγραμμα δεν είναι δυνατόν να μην μπορεί να εφαρμόσει το πρόγραμμα αυτό. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει το Συμβούλιο και το Συμβούλιο αποφασίζει για την πολιτική. Οπότε ένα βήμα θα μπορούσε να ήταν στη συνέχεια ο συνδυασμός ε, της θέσης του ε, Πρόεδρου της Επιτροπής και του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τουλάχιστον αυτός ο Πρόεδρος με το πολιτικό του πρόγραμμα θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στις ε, κατευθυντήριες ε, γραμμές ε, του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Έτσι θα είχαμε κάποια διαφορά. Μικρή βέβαια. Αχ, δυστυχώς έχω μακρηγορήσει. Θα βιαστώ προς το τέλος. Οικονομική και δημοσιονομική πολιτική. Αυτές περιλαμβάνονται στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε τέτοια περίπτωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια των νέων της λειτουργιών με το νέο σύστημα θα είχαν περισσότερο νόημα και θα είχε διαφορά αν ο πρόεδρος της Επιτροπής ε, είναι σοσιαλιστής και μια σοσιαλιστική πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα ήταν ε, επίσης διαφορετικό αν ήταν συντηρητικός ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η πλειοψηφία η κρατούσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αυτό θα άλλαζε τη φύση του προγράμματο και αυ, θα είχε νόημα και για τον κόσμο, ανάλογα με το τι δημοσιονομική πολιτική και τι πλαίσιο δημιουργείται. Βέβαια δεν έχουμε φτάσει ακόμη εκεί, έχουμε πολλά βήματα ακόμη για να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση και κάτι τέτοιο προποθέτει μια αναθεώρηση τη συνθήκης. Και δεν είμαι βέβαιος ότι η Βρετανική κυβέρνηση, η Μεγάλη Βρετανία θα συμφωνούσε σε μια τέτοια αναθεώρηση της συνθήκης. Πάντως αν κάτι τέτοια φορά μόνο τις χώρες Ευρωζώνης ή μόνο τις 25 από τις 27 χώρες, τότε ίσως ευοδοθεί μια τέτοια αναθεώρηση της συνθήκης. Και έρχομαι στο τελευταίο σημείο, τα διάφορα οράματα και τον πολιτικό μεσιανισμό. Νομίζω ότι υπήρξε ομοφωνία ότι η καλύτερη επιλογή εξακολουθεί να παραμένει μια ενιαία ενωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μια Ευρώπη πολλών ταχυτήτων αλλά ένωση κρατών εθνών. Οπότε η, η ομόφωνη λύση μάλλον φαίνεται να είναι η ενότητα. Και ίσως καλό θα ήταν να ξεκινήσει πολύ γρήγορα μια συζήτηση για το τι αντιπροσωπεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι εξυπηρετεί, για ποιο λόγο υπάρχει. Μερικοί πολιτικοί, πολιτικοί ηγέτες, ε, το αναφέρουν και ακόμη και στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια εξετάζεται μερικές φορές, αλλά δεν έχει γενικευτεί αυτή η συζήτηση στα κράτη-μέλη. Και ανάλογα με την έκβαση αυτής της συζήτησης, και άσχετα με την έκβαση συζήτηση, σίγουρα τη χρειαζόμαστε για να μπει αυτό το θέμα στην καθημερινότητα, να μπει επιτάπητος σε συνδυασμό και με το νέο σύστημα και με τις νέες εκλογές. Είναι σημαντικό να γίνει τέτοια συζήτηση γιατί ε, ενισχύει και την αίσθηση του κόσμου ότι βρίσκεται σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση, άσχετα με το τι μορφή θα έχει αυτή. Άσχετα με θα είναι ομόσπονδη, διεθνή οργάνωση, η Ένωση. Το θέμα είναι τι, τι σημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι εξυπηρετεί. Το θέμα είναι να είναι ένα καλό όργανο, ένα καλό εργαλείο για τις ευρωπαϊκές χώρες να συμμετέχουν στην διαμόρφωση των πολιτικών και να ανακτήσουν πολιτικές, την πολιτική του ισχύ στις χρηματαγορές. Αντί να περιμένουν από τις χρηματαγορές να μας βοηθήσουν να εξέλθουμε από την κρίση. Γιατί γνωρίζετε με το σύστημα της ΟΝΕ 121 άρθρα 121-126 στηρίζονται στην ε, υπόθεση α, ότι αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δώσει κίτρινη κόκκινη κάρτα σε ένα α, κράτος ότι δεν τα πάει καλά στη, στις α, ε, πολιτικές, στις οικονομικές, αντιδρούν οι αγορές και τιμωρούν ουσιαστικά το κράτος. Αλλά αυτό δεν το έκαναν οι χρηματαγορές ουσιαστικά. Η προσέγγιση ήταν ασφαλμένη. Και περιμέναμε από τις χρηματαγορές να μας βοηθήσουν και από τη δική τους δύναμη. Υπολογίσαμε στη δική τους δύναμη. Τώρα αντίθετα θα πρέπει να αναπτύξουμε τη δική μας ισχύ και να ανακτήσουμε την δύναμη που αφήσαμε στις χρηματαγορές. Και ίσως αυτό θα μπορούσε να είναι και ένα μήνυμα προς τον λαό, στον κόσμο, σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο, για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέες μορφές συμμετοχής ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το επισήμανε νομίζω ο Άντριο Ντάφ. η Μεγάλη Βρετανία και η Τουρκία συνδεθούν με κάποιο τρόπο. Και ορισμένα, με ορισμένα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ίσως αυτό θα ήταν μια απειλή προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Που αν υλοποιηθεί, φαντάζομαι θα εσπεύσει το Ηνωμένο Βασίλειο και θα συμφωνήσει απαραίτητε αναθεωρήσει και αλλαγέ τη συνθήκη για να έχουμε μία λειτουργική υγιή οικονομική και νομισματική ένωση και μια καταπληκτική Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά. Λίγα λεπτά έχουμε ακόμα. Το λόγο ζήτησε ο κύριος Νταφ. Για σύντομη ερώτηση και μετά θα μπορέσει να απαντήσει μόνο ένας από τους ε, ε, εμπειρογνώμονές μας και ε, θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Τσαρκόφσκι για να ε, κλείσει. Ο κύριος Νταφ. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω, Πρόεδρε, όλους τους ομιλητές μας και να πω ότι εκτιμήσαμε πάρα πολύ όλοι οι παρόντες στα λεγόμενά τους. Παρ' όλα αυτά, εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι να βρούμε έναν τρόπο να σχεδιάσουμε κάτι, εν περιπτώσει, που να ονομάζεται κυβέρνηση. Όχι διακυβέρνηση, κυβέρνηση με υπουργούς και υπαλλήλου που να ε, λειτουργεί ως κυβέρνηση, ως περιμένουμε εμείς ε, από τις κυβερνήσεις να δρουν. Αλλά μέχρι να φτάσουμε ως εκεί και πριν έχουμε μια ουσιαστική κυβέρνηση δεν πρόκειται να υπάρχει κοινοβούλιο που να αναγνωρίζει ο κόσμος ως γνήσιο και πραγματικό κοινοβούλιο, το οποίο να δρά όπως περιμένει ο κόσμος να δρουν τα κοινοβούλια. Και τώρα που τελειώνει αυτή η ακρόαση, θα ήθελα να έχουμε έτσι μία ενθάρρυνση να σκεφτούμε τι θέλουμε να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι σε αυτή την κυβέρνηση και που δεν γίνεται σήμερα. Χρειαζόμαστε μια κυβέρνηση που θα ασκεί ας πούμε βιομηχανική πολιτική. Όχι μόνο δάνεια. Θέλουμε κάτι που να είναι γνήσια δημοσιονομική πολιτική όχι μόνο δαπάνες, αλλά και τα έσοδα να κοιτάει. Επίσης, χρειαζόμαστε κάτι που να ε, ασκεί κοινή οικονομική πολιτική, όχι απλώς να συντονίζει εθνικές οικονομικές πολιτικές. Και επίσης κάτι άλλο που χρειαζόμαστε, και ίσως αυτό είναι το σημαντικότερο το τελευταίο που λέω, είναι Μία κυβέρνηση που να ασκεί δημοκρατική πολιτική. Τι εννοώ. Δεν ομιλώ μόνο για ε, τη διακυβερνητική ή διαθεσμική μάλλον ισορροπία ε, δυνάμεων ή μια ρητορική δέσμευση θεωρητική ε, σε δημοκρατικές αρχές. Αλλά ένα μόρφωμα που να λαμβάνει σοβαρά υπόψη την αναδυόμενη μετακρατική διάσταση ε, της ευρωπαϊκής πολιτικής. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν θέλει κανείς να απαντήσει. Δεν έχουμε πολύ χρόνο μετά από αυτό που πρότεινε ο κύριος Δαφ, θέλετε να σχολιάσετε ίσως. Όχι. Αν θέλει να ζητήσει κανείς το λόγο πρέπει να το κάνει τώρα. Όχι. Αλλιώς ε, να δώσουμε το λόγο στον συνάδελφο Τσαρκόφσκι για να κλείσει, να μας παρουσιάσει τη σύνθεση και τα συμπεράσματα από πλευράς ε, Κοινοβουλίου και Συνταγματικής Επιτροπής. Παρακαλώ. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή ε, κατάληξη και συμπέρασμα από τον καθηγητή Περνής και θα ήταν εκ μου ίσως ε, απρεπές να ε, κάνω μια σύνοψη τα συμπεράσματα. Απλώς να αναφέρω μερικά επιγραμματικά. Ε, όλοι ομολογούμε ότι λίγο μας ξεπερνούν οι εξελίξεις, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε διαπραγματευόμαστε και με τα άλλα θεσμικά όργανα. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα να προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες που είναι εγγενείς στις συνθήκες. Μετά, να προσπαθήσουμε να διαφυλάξουμε τη μοναδικότητα του ευρωπαϊκού μας εγχειρήματο, γιατί εκεί είναι πραγματικά η μεγαλύτερη ισχύ μας παρά τις όποιες δυσκολίες. Και ε, σε αυτή τη διαδικασία να προσπαθήσουμε να ε, υπερασπίσουμε την ακαιρεότητα των θεσμικών μας οργάνων. Ακούσαμε ότι αυτό δεν θα είναι εύκολο. Θέλουμε ε, ε, ευέλικτες λύσεις, πολυεπίπεδες, χωρίς να διαφυλαχθεί η ενότητά μας και ιδιαίτερα η ενότητα στο στόχο. Για το μεσιανισμό, δεν το έχουμε αυτό στην πολωνική ρομαντική μας παράδοση του 19ου αιώνα, όπου υποτίθεται ότι ήμασταν ο Μεσσίας της Ευρώπης. Και αυτό βέβαια μετριάστηκε από δύο αυταρχικά καθεστώτα και ε, αρχικά και ολοκληρωτικά και καθυστέρησε. Ε, συμφωνούμε για πολλές ε, λύσεις, αλλά θα πρέπει να υπάρχει περισσότερη ορατότητα, περισσότερη προβολή και για τον κόσμο και για τις επιλογές που ανοίγονται και χάρηκα πολύ που άκουσα τις ενδιαφέρουσες συνταγές σας. Όλοι έκαναν παραθέσεις. Να σας πω και εγώ την αγαπημένη μου από τον Μάρκ Τουέιν. Όταν βρίσκεσαι ε, στην πλευρά της πλειοψηφίας έχει έρθει η ώρα να κάνεις ε, μια στάση και να σκεφτείς και να προβληματιστείς. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Ε, σας διαβεβαιώ ότι ε, όλα αυτά που μας είπατε θα τα σκεφτούμε, θα προβληματιστούμε και θα συνεχίσουμε. Ευχαριστώ και εγώ, λέει ο Πρόεδρος. Ε, όλους προσκεκλημένους. Για μένα προσωπικά ήταν πάρα πολύ ε, ενθαρρυντικό ε, αυτό το σεμινάριο. Μου έδωσε μεγάλη τροφή για σκέψη, θα ευαθύνουμε, αλλά μου φαίνεται ότι ήταν πάρα πολύ σημαντική η συνεισφορά σας και σας ευχαριστώ. Και στο επανειδύνα. Possiamo togliere la seduta. Λίγεται η